Okay, Ωραία, πέρασαν αυτά τα λεπτά. Ήρθαν και οι σκιώδεις. Όχι όλοι, αλλά τέλος πάντων. Θα αρχίσουμε. Θα δώσω το λόγο στην Μόικα Κλέβα Κέκουσου που είναι η συγγήτρια, είναι εφαρμογή και αντίκτυπο των μέτρων ενεργειακή απόδοσης στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Έχω την εντύπωση ότι θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε μπροστά σας ένα σύντομο έγγραφο εργασίας που θα αποτελέσει τη βάση της μελλοντικής μου έκθεσης. Θα χαρώ πολύ να ακούσω τις δικές σας απόψεις γιατί αυτό θα με βοηθούσε στη συγγραφή της έκθεσης σύμφωνα βέβαια με τη γραμμή που έχει χαράξει η Επιτροπή μας. Η ενεργειακή αποδοτικότητα βρίσκεται στην καρδιά της στρατηγικής μας για βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε αναγνωρίσει ότι είναι κάτι πολύ θετικό, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά για να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης κατά 20%, της εξοικονόμησης κατά 20% της ενέργειας. Επομένως, πρέπει να καταλάβουμε ότι η σημασία που έχει η μεγαλύτερη και περισσότερη αποδοτικότητα και για την καταπολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών. Η επένδυση στην ενεργειακή αποδοτικότητα θα μπορούσε να καταλήξει σε απτά και άμεσα αποτελέσματα και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη μείωση του κόστους, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. και οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου. Επειδή η πολιτική συνοχής δε είναι από τα τμήματα της πολιτικής που μπορεί να πετύχει αυτόν τον στόχο, η Κομισιόν σκοπεύει στην επόμενη προγραμματική της περίοδο να διπλασιάσει σχεδόν το ποσοστό του προϋπολογισμού που αφιερώνεται στην πολιτική συνοχή. Δηλαδή αύξηση της χρηματοδότησης για προγράμματα μεγαλύτερης ενεργειακής αποδοτικότητας υψηλότερο προϋπολογισμό τους, ισχυρότερη θέση τους με τη σύγκριση με άλλα προγράμματα και σαφέστερο ρόλο της ε, στρατηγικής οικονομικής αποδοτικότητας. Αυτά είναι τα τρία θεμέλια της μελλοντική μας στρατηγικής. Οι διαπραγματεύσεις για το πολιετές πλαίσιο του προϋπολογισμού, πολιετή χαρακτήρα, ακόμη δεν έχουν τελειώσει. Αλλά καλό θα ήταν να υπενθυμίσουμε στα κράτη-μέλη ότι μια πολιτική συνοχή με σωστή χρηματοδότηση είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί αν δεν υπάρχουν οι χρηματοδοτικές δεσμεύσεις δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους τη στρατηγικής του 2020. Με την έκθεσή μου λοιπόν θα ήθελα να συμβάλλω και εγώ στη συζήτηση για την ενεργειακή απαδατικότητα μέσω της λήψης συγκεκριμένων μέτρων και της πρότασης ορισμένων από αυτά τα επόμενα χρόνια. Δεν θα ήθελα όμως να ανακατευτώ με την εντολή που δώσαμε το καλοκαίρι στους συναδέλφους <clears throat> όταν ψηφίσαμε για ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο για την Πολιτική συνοχή και όταν εγκρίναμε συγκεκριμένους κανονισμούς για συγκεκριμένα ταμεία. Θέλω αντίθετα την κοινοβουλευτική μας συζήτηση να τη χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουν τα θεσμικά όργανα εδώ στις Βρυξέλλες και εθνικοί οργανισμοί, τοπικές αρχές, περιφερειακές αρχές να διαθέτουν μία σαφή ανάλυση της κατάστασης, της ισχύουσας κατάστασης, ώστε να μπορούν να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Θα ήθελα στην έκθεσή μου να ασχοληθώ με τρία κύρια θέματα. <clears throat> την επιτυχή εφαρμογή καταρχήν των ήδη εγκεκριμένων μέτρων. Να δούμε γιατί έχουν, α και αν έχουν πετύχει και να διατυπώσω προτάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα πλαίσια πάντα της πολιτικής συνοχής. Η έκθεση φυσικά θα βασίζεται και στην πολιτική της στέγασης και του οικοδομικού τομέα γενικότερα. Γιατί εκεί υπάρχει το η μεγαλύτερη δυνατότητα εξοικονομήσεων. Πρέπει να αρχίσουμε από τα κτίρια νομίζω. Και πέρα από αυτό όμως δεν θα αγνοήσω ούτε παραγνωρίσω άλλους τομείς ενωσιακής και περιφερειακής οικονομίας που έχουν επιπτώσει στην ενεργειακή αποδοτικότητα όπως οι δημόσιες μεταφορές, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι υποδομές, οι ενεργειακές υποδομές και η αποθήκευση ενέργεια κλπ. Όταν αναλύουμε τα μέτρα λοιπόν ενεργειακής αποδοτικότητας θα ήθελα να απομακρυνθούμε από τις λεγόμενες ρυθμιστικές διαστάσεις και να βασιστούμε στις βέλτιστες πρακτικές και στα προβλήματα που μπορεί να ταυτίσουμε. Στην τελευταία έκθεση της Προεδρίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου κατέληξε ότι οι παράγοντες που καταλήγουν σε σπατάλη της ενέργειας πρέπει να αντιμετωπιστούν πρακτικά και όχι αφηρημένα και θεωρητικά. Όπως παραδείγματος χάρη να τεθεί το θέμα της ανεπαρκούς εφαρμογής της ισχύουσας ήδη νομοθεσίας. Επομένως, πέρα από τη λήψη νέων μέτρων όπως την οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα και για τα κτίρια, θα βασιστώ και στην τελευταία έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που μιλάει και για την αποδοτικότητα της ενέργειας. Επίσης ελπίζω πληροφορίες να πάρω και από την προεπικείμενη στρατηγική έκθεση της Κομισιόν για την εφαρμογή των προγραμμάτων 7 με 13 που θα δημοσιευτεί τώρα τον Μάρτιο. Τέλος, θα ήθελα να μιλήσουμε και για το μέλλον, δηλαδή κυρίως δύο στοιχεία. Πρώτον, σχεδιασμός και σύλληψη των μελλοντικών μέτρων και δεύτερον οι απαραίτητες ρυθμιστικές νομοθετικές αλλαγές ανάλογα με τα διάφορα κυβερνητικά και διαχειριστικά επίπεδα και συνδυασμό των διαφόρων ταμείων. Έτσι νομίζω η έκθεσή μας θα εισακουστεί. Γνωρίζω πολύ καλά τι δουλειά έχει κάνει η Επιτροπή μας ως πως τον γενικό κανονισμό του συγκεκριμένους για τα μεμονωμένα ταμεία δεν θέλω να υπάρξει καμία επικάλυψη ούτε επιχειρημάτων ούτε μέτρων αλλά να μιλήσουμε για τα καινούργια μονοθέματα και γι' αυτό θα περιορίσω την έκθεσή μου σε ό,τι αφορά αποκλειστικά και μόνο την ενεργειακή αποδοτικότητα. Θα ακούσω με χαρά τις ιδέες σας και τα σχόλιά σας και γνωρίζω πολύ καλά ότι θα συνεργαστούμε για να είναι η έκθεση πολύ στεναρή και να ακουστεί και από τους άλλους. Σας ευχαριστώ. Η η κυρία και παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε πρέπει να πω ότι είναι πραγματικά πολύ πλήρη η παρέμβαση. Ευχαριστώ ε, την εισηγήτρια για αυτό το σχέδιο έκθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη. Πρέπει να σα πω εξ αρχή ότι έχω την εντύπωση ενό δεζαβή πριν δύο εβδομάδε ε, συζητήσαμε το ίδιο θέμα. Μάλιστα ψηφίσαμε την ενεργειακή αποδοτικότητα στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχή και δύο μήνε μετά Μόλις έχουμε το ίδιο θέμα, κάπως πιο περιορισμένο βέβαια, γιατί στην έκθεση αυτή μιλάμε μόνο για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Όμως νομίζω ότι τίθεται το θέμα να ρωτήσουμε αν χρειαζόμαστε δύο εκθέσεις ουσιαστικά επάνω στο ίδιο ζήτημα. Γιατί όπως ε, υπόθηκε, παρουσιάστηκε με πολύ ενδιαφέρον τρόπο αυτό το θέμα. Ως και όδες εγώ θα υποστηρίξω την ανάπτυξη του θέματος αυτού, γιατί εγώ θεωρώ ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι ζωτική σημασία και αυτό αναγνωρίστηκε και στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Θα ήθελα η έκθεση αυτή να επικεντρωθεί κυρίως στον τομέα της κατασκευής κτηρίων και κατοικιών, αλλά και δημόσιων κτηρίων. Γιατί στον τομέα αυτό έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε, υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια και πάρα πολλά σπίτια που δεν σέβονται τα πρότυπα των, της καλής συνεργειακής απόδοσης. Εμείς θεωρούμε ότι το να θέσουμε πιο φιλόδοξους στόχους δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Επομένως, εμείς δεν ταχθούμε σε κάτι τέτοιο. Μάλιστα, θέτουμε το ερώτημα αν έχει νόημα να μεταφέρουμε πόρους από τη γραμμή του προπολογισμού που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προς την ενεργειακή αποδοτικότητα. Πραγματικά αναρωτιόμαστε αν κάτι τέτοιο θα είχε νόημα και κυρίως ε, είμαστε κατά του να πάρουμε πόρους από το μισονοχής και να τα μεταφέρουμε στον τομέα της ενέργειας. Όλα αυτά είναι μια καινοτομία. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο από του υπόλοιπου και συζητητέ. Ε, ίσως βέβαια να υπάρχουν εδώ κάποιοι συνάδελφοι που θα ήθελαν το λόγο να μιλήσουν για το έγγραφο εργασία. Στρέφουμε και στου εκπροσώπου τη Κομισιόν. Υπάρχει κάποιος που θα θέλει να αντιδράσει. Παρακαλώ. Σας δώσω το λόγο. Πώς μπορείτε να μας πείτε και πώς λέγεστε. Μάλιστα, σε ευχαριστώ. Είμαι από τη Γενική Διευθυνσή για την ε, αστική και περιφερειακή πολιτική της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ για τη δουλειά σας. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη και έρχεται την κατάλληλη χρονική στιγμή. Αυτός ο τομέας έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία τα τελευταία χρόνια με τους στόχους για το 2020, για την ενεργειακή εξοικονόμηση, και με την αναδιατύπωση της οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων και με την οδηγία για την νέα ενεργειακή αποδοτικότητα. Έχει συμμετέχει σε όλα αυτά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βλέπουμε πόσο αυξάνεται η σημασία των θεμάτων αυτών ε, στα σημερινά προγράμματα πολιτικής συνοχής. Έχουμε και αύξηση του προπολογισμού. Στο παρελθόν είχα 4 δισεκατομμύρια για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σήμερα μιλάμε για 5,5 εκατομμύρια που έχουν προβλεφθεί, δισεκατομμύρια με που έχουν προβλεφθεί. Έτσι λοιπόν βλέπουμε να αλλάζουν οι προτεραιότητες στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες. Και χάρη σε αυτή την τροπολογία που αναφέρθηκε, που έγινε το 2009, έχουμε και επιλεξιμότητα για επενδύσεις ε, σε κατοικίες σε όλα τα κράτη-μέλη. Όπως ακούσαμε λοιπόν, προτείναμε και τώρα διαπραγματευόμαστε μαζί σας στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το πλαίσιο για το επόμενο περίοδο. Προτείναμε να, να εστιάσουμε σε αυτό το τομέα, όπως αναφέρθηκε, με τις ελάχιστες ε, κατανομές ε, του προπολογισμού και φυσικά με αυτό το στόχο του 20% για την ενεργειακή αποδοτικότητα για το 2020. Και επίσης ε, προτείνουμε να εργαστούμε λιγότερο με επιδοτήσεις ε, και με περισσότερο με άλλα μέσα, όπως η χάρη εγγυήσεις δανειακές, για να έχουμε ένα αποτέλεσμα μόχλευσης και θα μπορέσουμε να έχουμε πολλά διδάγματα από τη σημερινή περίοδο. Επίσης, Πιστεύω ότι αυτός ο δικός χάρτης ε, που απαιτείται στην ε, νέα οδηγία ενεργειακής αποδοτικότητας και κάθε κράτος μέλος πρέπει να προετοιμάσει μέχρι του χρόνου τον Απρίλιο. Ε, ήδη ε, θα είναι πολύ, κάτι πολύ σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό έγγραφο από στρατηγική σκοπιά και θα μας βοηθήσει να καθοδηγήσουμε το σχεδιασμό των ε, επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η έκθεση αυτή λοιπόν θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Εξετάσαμε και τι έγινε το 2011. Κάναμε μια αξιολόγηση για το τι έκαναν τα κράτη-μέλη σε σχέση με την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις κατοικίες, ε, όμως ε, ήταν κάπως νωρίς. Έτσι λοιπόν, τώρα μπορείτε να δείτε κάποια καλά παραδείγματα και αυτό θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όλα τα κράτη-μέλη όταν θα προετοιμαστούν για την επόμενη περίοδο. Και επίσης πολύ χρήσιμα θα είναι και συστάσεις που μπορείτε να διατυπώσετε. Επίσης πρέπει να έχουμε κατά νου ότι διαφέρει η κατάσταση από κράτο μέλο σε κράτο και από περιφέρεια σε περιφέρεια και κυρίω σε ό,τι αφορά σε κτίρια κατοικιών όπου έχουμε διαφορετικέ συνθήκε. Πάντοτε θα ε, υπάρχουν κάποια μέτρα που θα αποφασίζονται ανάλογα και με τη συγκεκριμένη κατάσταση. Έτσι λοιπόν οι συστάσεις και καλές πρακτικές είναι όλα αυτά πάρα πολύ χρήσιμα. Και ας μην ξεχνάμε ότι θα χρειαστεί να υπάρχουν και συγκεκριμένα μέτρα για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δύο παρατηρήσεις μπορώ να κάνω εγώ. Καταρχήν, όσον αφορά την ε, ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση, ιδιαίτερα αν κοιτάξουμε τα μέσα συνοχής, ίσως θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο την αλλαγή που έγινε το 2009 του κανονισμού. Αυτή τη στιγμή το κείμενό σας ε, λέει ότι ήταν ε, μια πρόσθετη αλλαγή, αλλά ουσιαστικά ήταν μια μεγάλη αλλαγή. Είπατε ότι θα εξετάσετε κυρίως ε, τις καλές πρακτικές. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω ποιες ήταν οι κακές πρακτικές, γιατί δεν υιοθετήθηκαν όλα αυτά. Στο επόμενο διάστημα θα έχουμε και πάλι αυτές τις δυνατότητες χωρίς να έχουμε υποχρεωτικό στόχο για την ενεργειακή απόδοση. Θα είναι λοιπόν ε, σημαντικό να γνωρίζουμε γιατί σε κάποιες περιπτώσεις έγινε και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όχι. Ίσως θα μπορούσα λοιπόν να ζητήσω στην έκθεσή σας να έχετε μία ε, κύρια παράγραφο για το θέμα αυτό. Διότι εμείς ε, αυτό αλλάξαμε στον κανονισμό και τώρα που ολοκληρώνουμε τη δουλειά μας πάνω στον νέο κανονισμό με βάση την εντολή. Μας ενδιαφέρει και η εφαρμογή. Εκπρόσωπος της Κομισιόν ήδη είπε ότι υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις, διάφορες θέσεις στο θέμα της ενεργειακής απόδοσης. Η παρατήρησή μου είναι λοιπόν, παρακαλώ το θέμα της στέγασης να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο την έκθεση, της έκθεσής σας, ώστε να μπορέσουμε να καθορίσουμε τους στόχους της ε, περιφερειακής πολιτικής. Κοιτώ την αίθουσα, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε το λόγο κατευθείαν ε, στην εισηγητρία. Ναι, να, να πω λίγα λόγια τώρα στο τέλος. Ε, συμφωνώ με την κυρία Κολάσκα Πομπίνσκα και θα ήθελα να τη διαβεβαιώσω ότι ένα από τα σημαντικά θέματα της έκθεσης θα είναι ακριβώς ε, η στέγαση και οι οικοδομές. Ε, στην Επιτροπή Γυναικών ε, θα ψηφιστεί μια έκθεση για την κοινωνική στέγαση. Η Καρή επίσης συμμετέχει στις εργασίες, οπότε αυτό θα συμπεριληφθεί στην έκθεση αυτή. Όσον αφορά τις ευαίτησες πρακτικές, ε, συμφωνώ απόλυτα, είναι ενδιαφέρον ε, να δούμε γιατί είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα η εφαρμογή όταν μιλάμε για την ενεργειακή απόδοση. Θα προσπαθήσω λοιπόν να εντοπίσω, δεν θα έλεγα τις κακές πρακτικές, αλλά να επικεντρωθώ στο γιατί δεν εφαρμόστηκαν τα όσα συμφωνήθηκαν. Συμφωνώ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την προσπάθεια να προωθηθούν τα σχετικά οικονομικά μέσα. Ε, υποστηρίζω λοιπόν ε, τη χρήση ε, ε, την εφαρμογή των οικονομικών μέσων. Ε, πρόκειται για ένα έγγραφο εργασίας αυτό που είδατε. Προσπάθησα να βάλω κάποιες ιδέες, να καταγράψω κάποιες ιδέες. Η έκθεση θα εκπονηθεί ε, μέσα στις επόμενες εβδομάδες ε, και θα συζητηθεί στην Επιτροπή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις παρατηρήσεις σας. Ε, θα τις λάβω υπόψη μου κατά τη συγγραφή της έκθεσης. Ευχαριστώ. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση αυτή. Και τώρα διακόπτουμε μέχρι τις 10. Έτσι δεν είναι. Μισή ώρα διακοπή. Πρώτη μου φορά καθόμουν εδώ πέρα και ε, τα ολοκληρώσα μέσα σε μισή ώρα. Πρόκειται για μια τάση. Μπορείτε να μας πείτε ιστορίες από την παιδική σας ή κάτι τέτοιο, άμα θέλετε. We prefer the political career. <laughs> Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ ας ελέγξουμε τα μηχανήματα. Ε, θα κάνουμε λοιπόν την δοκιμαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Είμαστε λίγοι. Έχουμε απαρτία όμως. Κάποιοι δεν ψήφισαν. Δεν ξέρω μήπως δεν λειτουργούν οι συσκευέ. Ε, μόνο 26 φαίνεται να ψήφισαν. Λήξη τη ψηφοφορία. Από ό,τι κατάλαβα δεν υπάρχει πρόβλημα. Κωνσταντζα παρακαλώ. Πρωτού να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία της έκθεσης ο Μαρζή. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και μια παρατήρηση. Καταρχήν να πω ότι η πολιτική μας ομάδα με κανένα τρόπο δεν είναι κατά ε, της ε, βοήθειας, ε, βοήθειας προς τους στοχότερους της Ευρώπης. Αλλά έχουμε ε, κάποιες δυσκολίες με την έκθεση. Στην αρχή υπήρχε μόνο στα γαλλικά. Έχω αναφέρει τις δυσκολίες. Ε, τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο της ψηφοφορίας ε, και διαπιστώνω ότι δύο πράγματα είναι προβληματικά στη γνωμοδότηση αυτή. Καταρχήν το θέμα της αύξησης ε, του προϋπολογισμού των πόρων. Η ε, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ε, στο, στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπουν μείωση και εδώ πέρα. Είχαμε τον, κανον, τον κανόνα να αφήνουμε ε, εκκρεμές το θέμα αυτό και τώρα βρισκόμαστε ε, προ ψηφοφορίας για τον προϋπολογισμό. δεν μπορούμε εν μέσω διαπραγμάτευσης να εγκαταλείψουμε τις διαπραγματεύσεις ε, και να υπερψηφίσουμε μια αύξηση. Επίσης ε, υπάρχουν εδώ πολλές τροπολογίες που έχουν να κάνουν με το σύστημα ελέγχου και διαχείρισης από πλευράς της Κομισιόν. Μάλλον θέλουν να καταργήσουν το σύστημα αυτό. Ε, η πολιτική μας ομάδα θεωρεί ότι αυτό είναι κατά του δημοσιονομικού κανονισμού. Υπάρχει εκεί νέα νομική βάση. Η επισητιστική βοήθεια εμπίπτει στο κοινωνικό ταμείο και την πολιτική συνοχή. Είναι θέμα μοιρασμένης αρμοδιότητας και γι' αυτό θα πρέπει σε όλα τα επίπεδα να υπάρχει σχετικό σύστημα ελέγχου. Μπορούμε να συζητήσουμε αν θέλουμε ένα απλοποιημένο σύστημα στην περίπτωση αυτή, αλλά κατά τη γνώμη μας δεν μπορούμε να ε, το διαγράψουμε αυτό. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να αναβληθεί η ψηφοφορία, να ελεγχθούν τα θέματα αυτά. και να μπορέσουν να υποβληθούν νέες τροπολογίες και να βρεθούν νέοι συμβιβασμοί. Εάν δεν υπάρχει πλειοψηφία υπέρ της πρότασης αυτής και ψηφίσουμε, ε, παρακαλώ να σημειωθούν στο, ε, στα πρακτικά αυτά που είπα και να το θεωρήσετε και επεξήγηση ψήφου γιατί η ομάδα μας δεν μπορεί να υπερψηφίσει ε, την πρόταση. Ο κύριος Κάντεκ, παρακαλώ. Η μας εξηγεί γιατί δεν θέλει να ψηφίσει ένα τμήμα της έκθεσης αυτής, λέγοντάς μας ότι δεν είναι αντίθετη στην βοήθεια στους απόρους. Θεωρώντας ότι είναι υποσυζήτηση ο προπολογισμό, ε, δεν έχουμε αποφασίσει τίποτα ακόμα, αλλά κανείς εδώ δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι Ακριβώς στο πλαίσιο της κρίσης οι άποροι ε, δεν ε, περίμεναν καμιά άλλη στιγμή τόσο πολύ την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο σήμερα. Εγώ νομίζω τώρα ότι τεχνικά επιχειρήματα ή άλλου είδους δεν ε, ανήκουν σε τέτοια συζήτηση και νομίζω ότι είναι κρίμα να στηριζόμαστε σε τέτοια επιχειρήματα για να μην ψηφίσουμε αυτή τη διάταξη. Αυτό θέλω να πω. Πρόεδρος, ε, θέλουμε να έχουμε τη συζήτηση και κατόπιν θα δώσω την, ε, το λόγο στον εισηγητή, ο κύριος Λάμπερτ. Αν επιτρέπετε, έχω κάπως ε, προβληματιστεί. Γιατί ένα λεπτό πριν την ψηφοφορία αρχίζουμε να σκεφτόμαστε αν έχει προετοιμαστεί καλά το έγγραφο ή όχι. Η οχι Για δικη μου εντύπωση είναι ότι είχε εκπονηθεί ορθά. Έχουμε ένα καλό κατάλογο ψηφοφορίων. Και αν για κάποιους λόγους η Επιτροπή θέλει να δώσει ένα μήνυμα, μπορούμε ίσως να το κάνουμε με έναν άλλο τρόπο. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο αλλά είναι πολύ μικρό το ποσό και θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία. Η δική μου πρόταση ήταν να ψηφίσουμε. Να μείνουμε στους προετοιμασμένους συμβασμούς και να τους υποδεχτούμε για να μην χάνουμε χρόνο. Πρόεδρος, παρακαλώ, εισηγητής. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πραγματικά με εκπλήσει μια τέτοια συζήτηση που λαμβάνει η χώρα λίγα λεπτά πριν την ψηφοφορία, αλλά τουλάχιστον ίσως εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις ε, θέσεις των μεν των δε. Δηλαδή, θέλω να χαιρετήσω τους ε, συμβιβασμούς ο οποίος κατέληξε σχεδόν το σύνολο των πολιτικών ομάδων και το έργο που υλοποιήσαμε για την εκπόνηση της έκθεσης αυτής. Τώρα, κάτι ακόμα τρίτο. Πιστεύω ότι οι βουλευτές που είναι παρόντες εδώ είναι ελεύθεροι να υπερασπίζουν τις θέσεις που θεωρούν σωστές. Ορισμένοι έχουν κάποιες απόψεις που έχουν συμπεριληφθεί στους συμβιβασμούς, ενώ κάποιες άλλες θέσεις είναι πιο προσωπικές και δεν υπάρχουν στους συμβιβασμούς. Σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό, το θέμα του προπολογισμού είναι μια συμβολική τροπολογία που εγώ θέλησα να καταθέσω προσωπικά, αλλά δεν αποτελεί μέρος των συμβιβασμών, δηλαδή ο καθένας είναι ελεύθερος να καθορίσει τη δική του θέση ανάλογα με όσα πιστεύει. Για το τελευταίο τώρα σημείο τέθηκε το θέμα στη γραμματεία της ε, Επιτροπής για το αν είναι αν ισχύουν ε, οι τροπολογίες ε, από νομική σκοπιά, απάντησε η Κομισιόν ότι ισχύουν και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να ψηφίσουμε, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια έκθεση την οποία την παραμένουν οι πολίτες. Έτσι λοιπόν δεν βλέπω εγώ λόγο να βολήσεις. Ευχαριστώ. Η Μαρή Τερές θέλει να πάρει το λόγο, αλλά δεν θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι κάναμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε στο δικό μας επίπεδο. Ε, δεν υπάρχει θέμα του απαράδεκτου, λέει η Γραμματεία. Σημειώνουμε τις παρατηρήσεις ε, της Κωνσταντσα. Δεν ξέρω αν το ίδιο ισχύει για τον ε, Λαμπέρ και τον Αλένα, αν θέλουν οι παρατηρήσεις τους να συμπεριληφθούν στα πρακτικά, αλλά αν το επιθυμούν μπορούμε να το κάνουμε. Θα ψηφίσουμε λοιπόν τώρα και μπορούμε να επιστήσουμε την προσοχή της Επιτροπής Απασχόλησης αν υπάρχει πρόβλημα. Ε, αν υπάρχει νομικό πρόβλημα, διότι ω επί τη ουσία αρμόδια επιτροπή μπορεί να αναλύσει περισσότερο ει βάθο το θέμα αυτό. Εάν δεν έχετε αντίρρηση λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Παρακαλώ. Πολύ σύντομα. Ε, μου φαίνεται ότι ξέχασα την κάρτα μου, αλλά θα ψηφίσω με το χέρι. Ωραία, η γραμματεία θα σας κοιτάει. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη συμβαστική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 152. Όχι. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε την 164, αρχή της ψηφοφορίας. 164 ψηφίζουμε. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 23 υπέρ, 16 κατά. Συμβαστική 5 υπέρ. 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρέπει να σταματήσω λίγο. Ε, so now we go to amendment 107. Προχωράμε στην 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 και 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 176-177 υπέρ κατά νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά να την ελέγξουμε. 176-177 Αρχή της ψηφοφορίας Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 20 υπέρ 20 κατά ε, απορρίπτεται και πάλι. 38 υπέρ κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται να ελέγξουμε γρήγορα την 38. Λήξη της ψηφοφορίας. <laughs> 20, ψήφοι υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές. Ε, νομίζω ότι έχουμε την πλειοψηφία, να την ελέγξουμε όμως, ε, διότι δεν το βλέπω. 39 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 22 υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται. Υπάρχει η προφορική τροπολογία για την ε, τροπολογία 40. Είναι κανεί κατά, ε, αλλιώς ψηφίσουμε υπέρ, κατά να ελέγξουμε την 40 όπως έχει τροποποιηθεί. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 22 υπέρ, 17 κατά, 178 ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 183. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 184. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 186. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ένα λεπτό. 189 και 188 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε τις 189 και 188. Λήξη της ψηφοφορίας. Πώς ψηφίσατε? Απορρίπτεται, απορρίπτεται. Η 45 καταπίπτει. δεν καταπίπτει. 45 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 190 και 191 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 193 και 192 είναι όμοιες υπέρ. Κατά να ελέγξουμε 193-192. Τις ελέγχουμε ηλεκτρονικά αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 47 και 194 είναι όμοιες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 48 και 196 ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 49 και 198, 199 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 201 και 200 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε τις 201 και 200. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Τι ψηφίστε κατά. Ε, απορρίπτεται λοιπόν 19 υπέρ 20 κατά. 50. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 50. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να το ελέγξουμε. Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 202 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 200... Η επόμενη καταπίπτει. Όχι, ψηφίζουμε τη 203 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 207 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 208 και 9 υπέρ. Κατά ελέγχουμε τις 208 και 209 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας Εγκρίνεται 23 ψήφοι υπέρ 17 κατά. Ένα λεπτό. Περιμένουμε. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μάλλον δεν είμαστε βέβαιοι, ελέγχουμε την 53. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 23 υπέρ, 16 κατά. 54 ε, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 213, όχι. 212, ψηφίζουμε 212. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 213, υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε τη 213. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 21 ψήφοι κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται ακόμα και αν ε, ψηφίσει υπέρ ε, η κυρία. Λοιπόν, 55 ε, υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε την 55 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 215 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε, συμβαστική ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 58. Υπάρχει προφορική τροπολογία, υπάρχει κανείς που να είναι κατά της προφορικής τροπολογίας, όχι, άρα ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 218 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 219 ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 221 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 222 και 223 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 224 και 25 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε, εγκρίνεται, συγγνώμη. 226 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. 227 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 228 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 229 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 229. αρχή της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 230 και 31. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 232 δεν την ψηφίζουμε. 242 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 233 και 234 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 235 και 236 υπέρ κατά ελέγχουμε 235 και 236 αρχή της ψηφοφορίας απορρίπτεται 17 υπέρ 22 κατά 237 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε τη 237 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 18 υπέρ 21 κατά. 59 υπέρ, ε, προφορική τροπολογία είναι κανείς κατά όχι. Ψηφίζουμε υπέρ. 59 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 60, καταπίπτει ή όχι. Ψηφίζουμε την 60, υπέρ, κατά, ελέγχουμε την 60. Λήξη της ψηφοφορίας. Ψηφίστε υπέρ ή κατά. Απορρίπτεται. 19 υπέρ, 20 κατά. 238 και 239 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. 238 και 239 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 20 υπέρ 18 κατά. Η 240 καταπίπτει. 61. Ψηφίζουμε υπέρ κατά να ελέγξουμε την 61 γιατί νομίζω ότι αλλάζουν οι συνασπισμοί ε, λήξη της ψηφοφορίας 20 υπέρ 18 κατά εγκρίνεται 241 ποιος είναι υπέρ κατά να ελέγξουμε την 241, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας, 21 ψήφοι υπέρ, 18 κατά. Ε, συμβαστική 14, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 249, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 248 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64 που τροπήθηκε κατά την μετάφραση. Ποιος είναι υπέρ. Της 64. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 251 και 252 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 255 υπέρ 255 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ένα λεπτό. So 72. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 72. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 260 και 61. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, ψηφίζουμε την 74. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 266 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 267 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίσουμε την 79. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 274, 75 και 76 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 80. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 80. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται 20 υπέρ 18 κατά 278 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 279 και 280 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ...283 και 284. Ποιος είναι υπέρ. 283-284 υπέρ, κατά. Ε, ε, ε, εγκρίνεται αν όλοι οι σοσιαλιστές σας ακολουθήσουν. Εγκρίνεται υπέρ. 285 και 286 υπέρ. Κατά. Πρέπει να την ελέγξουμε. Πολύ λίγοι από εσά πραγματικά ψηφίζετε. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 22 υπέρ 17 κατά εγκρίνεται. 58 or no, we'll go to in principle to 303. So we go now to 303. 303. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 304 είναι όμοια, συγγνώμη δεν το είπα. 305 υπέρ. Λαμπέρ, ποιο είναι υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 306 και 7, 306 και 7 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 308 και 9. Α, όχι, είναι όλε όμοιε. Ε, συγγνώμη. Ε, έχουμε ψηφίσει δηλαδή και την 311. Προχωράμε τώρα στην 312 και 313. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 314 και 315. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 316-317 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περιμένουμε ένα λεπτό, γιατί είναι πολύ πλοκά τα πράγματα. So we go now to 319. So we go to 319. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 320, 21 και 22. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. 320, 321, 322 και 323. The vote is closed and it is... Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 324 και 325. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 326 και 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 328 και 329 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 330 και 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 332 και 333 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 334 και 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 336 και 337 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 338 και 339 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 340-341 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 342 και 343 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 344 και 345 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 346 και 347 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 348 και 349 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 350 και 351 Α, συγγνώμη. Ε, βιάζομαι, μου φαίνεται. 350 λοιπόν μόνη της, ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 351 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 352 και 53 εγκρίνονται... Α, ε, ήδη έχουν υιοθετηθεί. Προχωράμε στα εκτιμώντας. Εκτιμώντας 1, τροπολογία 2, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 4, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 94, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική, ε, ε, τροπολογία 100 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να ελέγξουμε την 10. Την 10. Yeah, okay, maybe you're right, but we close the vote and it's 19 to... Λήξη της ψηφοφορίας, 19 υπέρ, 19 κατά. Α, όχι, εγκρίνεται διότι έχουμε 20 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. 101. 101 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εγώ βέβαια είμαι, αλλά σε ελέγξουμε. 110. Αρχή της ψηφοφορίας. Μόνο το ECR και οι σοσιαλιστές ήταν κατά. Εγκρίνεται 26 υπέρ, 14 κατά. 110 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ, κατά Να ελέγξουμε την 119. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 118 καταπίπτει. 120 ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε την 120. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται 121 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 29. Συμβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ κατά απορρίπτεται να ελέγξουμε την 129 αρχή της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται 19 υπέρ 21 ψηφί κατά 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 και 33 δεν τις ψηφίζουμε Δεν τις ψηφίσουμε. Προχωράμε στην 131, χωριστή ψηφοφορία. Ψηφίσουμε πρώτα το πρώτο μέρος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Όλα τα υπόλοιπα έχουν υιοθετηθεί, μου λένε εδώ. Προχωράμε στην 20 και την 145. Ε, Εκτιμώντα 27. Να με το λαμπέρ. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Είσαι κατά λαμπέρ. Ε, και αυτός είναι ρόλος μου. Δυστυχώς απορρίπτεται από ό,τι βλέπω. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. 23 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 147 και 148 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Και έτσι ολοκληρώσαμε. Εφτάσαμε στην τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 5 κατά, 9 αποχές. Εγκρίνεται. Okay. Uh, thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Προχωράμε στην επόμενη ψηφοφορία, κοινωνική στέγαση. By Monsieur Carona and who's helping me? it's okay. Fine. Thank you. Uh, can we start... Ο κύριος Καρανά, ο εισηγητής, να περάσουμε στο συνδεσμό ένα υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2. Υπέρ. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Αν δεν είναι κανείς κατά, ψηφίζουμε αυτό το συμβιβασμό όπως έχει τροποποιηθεί. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3. Συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27. Απολογή 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στο συμβολισμό 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5, συνδεσμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συνδεσμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 έχουμε δηματική ψηφοφορία το πρώτο τμήμα υπέρ κατά να ελέγξουμε για το πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία πέρας 23-17 εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Νομίζω απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε όμως γιατί δεν είμαι σίγουρη. Για το δεύτερο τμήμα παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Έχουμε 17 υπέρ 22 κατά 48. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Νομίζω απορρίπτεται, αλλά να ελέγξουμε. 48. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. 17-22. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. 36 υπέρ, καμία ψήφος κατά, τρεις αποχές. Σχεδόν τέλεια, συγχαρητήρια. Θα δοκιμάσουμε τις πληροφορίες. Παρακαλώ, Λέμπερ, να ανακοινώσω ότι υπάρχει μια μικρή μπροσούρα και αφορά την ευφύ εξειδίκευση και ξέρετε, εγώ θέλω να υπερασπιστώ αυτό το θέμα. Πάρτε αυτή την προσούρα. Είναι στα αγγλικά, δεν είναι στα ολλανδικά. Ειδικά για εσά. σα ευχαριστώ. sorry, but we... Θα διακόψουμε μέχρι να έρθει ο Επίτροπος. Ελπίζω ότι θα έρθει γέρος και θα συνεχίσουμε. Κύριε Επίτροπε, θέλουμε να αρχίσουμε. Uh, dear colleagues, we are... Αγαπητοί συνάδελφοι, ξαναρχίζουμε θα ζητήσω, θα δώσω μέσα το λόγο στον Επίτροπο να μας πει δύο λόγια και μετά οι ερωταπαντήσεις και τα σχόλια. Ορίστε κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ Ντανούτα. Ευχαριστώ Ντανούτα. Ζητώ συγγνώμη. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την δυνατότητα να ξαναβρεθώ εδώ πέρα για μια ανταλλαγή σχετικά με την κατάσταση μετά την συμφωνία τουλάχιστον σε επίπεδο κρατών μελών. Σας ε, ευχαριστώ πολύ ε, για την ε, οργάνωση αυτή του Κοινοβουλίου. Το θέμα είναι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των αγορών και των ιδιωτικών επενδυτών, ιδιαίτερα σε καιρούς όπως είναι οι παρόντες. Η πολιτική σημασία αυτού που αποφάσισαν τα κράτη-μέλη είναι πολλαπλή. Από τη μία έχουμε μία σαφή, ίσως όχι πολύ, σημαντική, πολύ μεγάλη αύξηση για την ε, έρευνα και την ανάπτυξη. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ε, ανεργία των νέων ε, από την άλλη όμως υπάρχουν και λιγότερα χρήματα για τις περιφέρειες ε, και τη γεωργία. Αλλά θα ήθελα εδώ να σημειώσω ότι ο προϋπολογισμός ανταποκρίνεται στη νέα αρχιτεκτονική της περιφερειακής πολιτικής. Σκεφτείτε για παράδειγμα την, ε, δημιουργία των ε, μεταπατικών περιφερειών και τις νέες στρατηγικές κατευθύνσεις της περιφερειακής πολιτικής. Δεν θα ήθελα να κρύψω ότι υπάρχουν σημεία που προσωπικά τα βλέπω με κριτικό μάτι. Ε, ε, εγώ και οι συνεργάτες μου μάλλον όμως είμαστε απομονωμένοι στο θέμα αυτό. Ε, να σκεφτούμε ότι ο κανόνας νη συν δεν έχει δημιουργηθεί για να δαπανούμε με καλύτερο τρόπο τα χρήματα, αλλά οδηγεί σε πολλές Ε, ε, αφορά πολλές προσπάθειες ε, των συνεργατών μου. Και μάλιστα ακυρώνει αυτές τις προσπάθειες των συνεργατών μου. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Με μια με ένα συντηρητικό υπολογισμό, τουλάχιστον το 40% του προϋπολογισμού που περιμέναμε, θα δοθεί μετά το 2020. Για να σας περιγράψω δηλαδή τι σημαίνει το νησιν 3. Επίσης ε, βρίσκω λυπηρό το ότι έχουμε περικοπές ε, στην εδαφική συνεργασία ε, που είναι ένας από τους τομείς ε, όπου είναι πιο ορατή η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι λάθος να στείλουμε ένα τέτοιο μήνυμα. Το Κοινοβούλιο κατά τις διαπραγματεύσεις, εάν θέλει να κάνει κάτι να βελτιώσει την κατάσταση, θα ήταν χρήσιμο να στείλει ένα σαφές ευρωπαϊκό μήνυμα παρά τις επικρίσεις, ε, τις οποίες ε, δεν θέλω να κρύψω. Η συμφωνία των ε, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων μπορεί να αποτελήσει χρήσιμη βάση για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Σημαντικό είναι να βρούμε μια γρήγορη λύση στο θέμα αυτό. Η περαιτέρω διαπραγματεύσεις προχωράνε και δεν θα πρέπει να μειώσουμε την ταχύτητα. Ε, είμαστε περήφανοι για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Ε, δεν θέλουμε να διακυβεύσουμε ε, έναν σίγουρο προγραμματισμό. Όλα τα κράτη-μέλη και τα μελλοντικά και η Κροατία δηλαδή έχουν κληθεί να υποβάλουν σχέδιο ε, συμφωνίας εταιρικής σχέσης, ώστε αμέσως ε, μόλις ε, ολοκληρώσουμε τα θέματα αυτά, να μπορέσουμε να ασχοληθούμε παράλληλα και με τα επιχειρησιακά προγράμματα. Θέλουμε λοιπόν μια ομαλή μετάβαση από τη μία περίοδο στην άλλη. Αλλά όπως σας είπα χρειάζονται και επίσημες αποφάσεις για, κάτι, για να συμβεί κάτι τέτοιο. Πολύ σημαντικό είναι να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε εξέταση τους δημοσιονομικού πλαισίου ε, που να ασχολείται με τα μεμονωμένα έτη μπορεί να διακυβεύσει την ε, περιφερειακή πολιτική, διότι η περιφερειακή πολιτική ε, βασίζεται στην ε, ασφάλεια προγραμματισμού, στην προβλεψιμότητα και στην βεβαιότητα όσον αφορά τους διαθέσιμους πόρους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο για τις προσπάθειές σας στον τρέχοντα τριμερή διάλογο. να ευχαριστήσω και τους εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές. Ε, νομίζω ότι όλοι μαζί κινούμαστε προς μια σωστή κατεύθυνση και πιστεύω ότι είναι ε, δικαιολογημένη η ελπίδα μέχρι το καλοκαίρι να έχουμε συμφωνία. Οι συνεργάτες μου και εγώ προσωπικά είμαι ανα πάσα στιγμή στη διάθεσή σας. Ε, δύο σημεία είναι σημαντικό να αναφερθούν. Ε, και που μπορούν να αποτελέσουν ε, αντικείμενο της σημερινή συζήτησης. Έχουμε αφενός ε, την συζήτηση για το ελάχιστο μερίδιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε φιλόδοξη λύση ώστε να βρούμε μια το ελάχιστο μερίδιο του ERDF και για να επιτρέψουμε την ε, απαραίτητη ευελιξία. Αλλά δεν θα πρέπει να αλλάξουμε την ε, βασική ιδέα. Δεύτερο θέμα, τώρα που μιλήσαμε για το better spending, για τον καλύτερο τρόπο να δαπανούμε τα χρήματα, μας ενδιαφέρει το θέμα ε, της θεματικής συγκέντρωσης. Παρακαλώ να μην δεχτείτε αποδυνάμωση στο θέμα αυτό, διότι εξυπηρετεί την εφαρμογή κοινών ευρωπαϊκών στόχων. Εάν δεν επικεντρωθούμε λοιπόν στους ε, στόχους αυτούς ε, και ε, διαθέσουμε τα, τους απαραίτητους πόρους, θα αποτύχουμε. Και ε, ιδιαίτερα σε χώρες ε, με λιγότερους πόρους εξασφαλίζεται η ορατότητα της Ευρώπης. Σημαντικό πάντως είναι να επικεντρωθούμε στα θέματα τα οποία θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε τους στόχους ε, του προγράμματος Ευρώπη 2020, τους στόχους ως προς την ανάπτυξη. Πιστεύω ότι η Κομισιόν έχει επιδείξει επαρκή ευελιξία, αλλά χρειάζεται ευελιξία από όλες τις πλευρές. Ε, ευελιξία όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ευελιξία σε όλα τα θέματα, διότι αυτό είναι παρερμηνία του όρου. Ε, χρειάζεται να έχουμε λύσεις ε, κομμένες ε, στα, μέτρα του καθενός. Ε, παρακαλώ λοιπόν να με στηρίξετε, διότι ξέρω ότι στις διάφορες εκλογικές περιφέρειες, στις περιφέρειες υπάρχουν ιδιαιτερότητες, αλλά μπορεί και είναι δυνατόν να επικεντρωθούμε στα θέματα αυτά που αποτελούν το περιεχόμενο της ε, στρατηγικής μας ε, για το 2020. Θα πρέπει να διαθέσουμε με ανάλογο τρόπο τους πόρους. Έτσι θα δημιουργήσουμε ε, Έτσι θα δημιουργήσουμε μια σωστή εικόνα της περιφερειακής πολιτικής αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Μας περιμένουν σκληροί μήνες. Ε, νομίζω όμως ότι τελικά... Ε, θα αξίζουν τον κόπο οι προσπάθειές μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας κατευχαριστώ Ιωάννη. αρχίσουμε με τους συντονιστάς. Υπάρχει πολύ μακρύς κατάλογος ομιλητών. Πρώτα όμως οι συντονιστές. Δεν θα ξεχάσουμε και τα απλά μέλη, μη φοβάστε. Λοιπόν, ο Λαμπέρ πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να είμαι σύντομος, γιατί τα συμπεράσματα από τους τριμερείς διαλόγους των τελευταίων μηνών είναι ότι η αρχιτεκτονική δομή της νέας πολιτικής συνοχής θα παραμείνει η ίδια. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Η νέα θεματική συγκέντρωση, τα κύρια θέματα δηλαδή, δεν είναι αμφιλεγόμενα. Αν το Κοινοβούλιο θέλει και το ICT, αυτό διότι έχει σοβαρό λόγο και το Συμβούλιο κάνει λάθος που το αρνείται. η Ευρώπη υποτίθεται ότι προετοιμάζει μια νέα εποχή νέες μορφές απασχόλησης, νέες μορφές δραστηριότητας και τι λέει, ζητάμε ένα δισεκατομμύριο. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι μια ένα συνδυασμό με το περιφερειακό και τοπικό δημοτικό επίπεδο. Διότι επανειλημμένος είπαμε ότι πρέπει να διευρυνθεί αυτή η παρατηρούμενη συγκέντρωση. Το έχουμε πει πολλές φορές και έχει αποδειχθεί ότι είχαμε δίκιο. Δεύτερον, το εξής. Λέτε ότι θα μπορούσαμε λίγο πριν ή λίγο μετά το καλοκαίρι να ληφθούν αποφάσεις. Ε, και εμείς αυτό θέλουμε. Και αυτό για όλους τους ενδιαφερόμενους στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αυτό περιμένουν όλοι. Αυτό θα ήταν μια συγκεκριμένη απάντηση, ανταπόκριση στην κρίση και δεν θα πρέπει να καθυστερήσουμε κι άλλο. Τώρα για το ΕΛΚ ειδικά επιμένουμε ιδιαίτερα σε αυτό να μην καθυστερήσει το πράγμα. Χαιρόμαστε πάντως που φαίνεται, διαφαίνεται κάποια λύση και κανονικά οι τριμερείς διάλογοι και τα κνακ πούγκτε όπως είπατε και εσείς, τα σημεία κλειδιά μπορούμε, τα σημεία τα αμφιλεγόμενα μπορούν να λυθούν. Τώρα, ερώτημα. Μετά το Συμβούλιο και τη Συμφωνία για το Πολδίπ δεν ξέρουμε ακόμη τι επιπτώσεις θα έχει αναχώρα δημοσιονομικά. Φαντάζομαι ότι εσείς το ξέρετε. Εμείς ακόμα δεν το μάθαμε. Θέλουμε να ξέρουμε αναταμείο και αναχώρα ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του Πολδίπ. Σας παρακαλώ λοιπόν να μας πείτε ό,τι ξέρετε, γιατί είναι δύσκολο να εργάζεται κανείς με βάση απλούς υπολογισμούς που μπορεί να αποδειχθούν και λανθασμένοι. Έπειτα, μιλήσατε για το κοινωνικό ταμείο. Πρέπει να σας πω ότι η Κομισιόν δεν κάνει τίποτα γι' αυτό συνολικά. Εσείς δεν ξέρω τι κάνετε το Συμβούλιο έλαβε θέση με συγκεκριμένα ποσοστά και εμεί επίση Η Κομισιόν τι κάνει, όμω, τίποτα. Αυτό νομίζω είναι ανεύθυνο. Μα είπατε πριν από λίγο ότι πρέπει να δούμε τα ποσοστά αυτά να είναι ευέλικτα και λογικά. Ναι, αλλά κάντε κάτι με τους άλλους επιτρόπους για να βρεθεί κάποιος συμβιβασμός. Ξέρω ότι και η Κωνσταντ θα σχολιάσει αυτό, γι' αυτό παραμένω σύντομος. Αλλά προσθέτω παρόλα αυτά το εξής. Όταν υπήρχαν δυσκολίες για το Connecting Europe, εμείς κάναμε τεράστια προσπάθεια για να βρούμε μια λύση. συνδυασμένη με το Ταμείο Συνοχής. Αν εσείς δεν κάνετε τίποτα για το Κοινωνικό Ταμείο, αν εσείς δεν προτείνετε τίποτα για να βγούμε από το αδιέξοδο, τότε ακόμα μια φορά το Κοινοβούλιο θα χρειαστεί να κάνει κάτι και μάλιστα μόνο του. Ευχαριστούμε η Κωνσταντς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Ε, δεν ε, θα πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία που έχουμε σήμερα που βρίσκεστε εδώ στην Επιτροπή μας ε, ώστε να έχουμε μια σαφή ανάλυση. Δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε την την πρόταση που υπάρχει, αλλά νομίζω ότι εάν δεν επιταχύνουμε στον τριμερή διάλογο, κινδυνεύουμε να μην ολοκληρώσουμε τις εργασίες μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και θα πρέπει να το πούμε αυτό σαφώς. Ε, τελευταία φορά που ήσασταν εδώ ε, νιώθαμε όλη η εφορία, ε, αισιοδοξία σχετικά με τα αποτελέσματα και πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο έχει κάνει αυτό που έπρεπε και όσον αφορά την προετοιμασία των θεμάτων με τη διαπραγματευτική μας ομάδα, με τον εισηγητή. Έχουμε υποβάλει προτάσεις, είμαστε διατεθειμένοι να βρούμε συμβιβασμό ε, υπάρχουν ελλείψεις όμως από την άλλη μεριά όσον αφορά το αποτέλεσμα. Να σας ε, αναφέρω παραδείγματα. Και μάλιστα δεν έχουμε καν ε, φτάσει ακόμα στα σημαντικά θέματα όπως είπε ο, Λάμπερτ. Δεν έχουμε συζητήσει το θέμα των μακροπρόθεσμων προϋποθέσεων. δεν μιλάμε για συμβασμό να, ε, για να συνενώσουμε τα δύο άκρα. Συζητάμε εν μέρη εάν τα κράτη-μέλη είναι διατεθειμένα όχι μόνο να ε, ε, προτείνουν, αλλά και να χρησιμοποιήσουν την ε, ηλεκτρονική συνοχή. Ώρες συζητάμε για αυτά τα θέματα και αυτό δεν οφείλεται στη δική μας πλευρά. Θέλω να το πω αυτό σαφώς. Πρέπει να επιταχυνθούν τα πράγματα και κυρίως πιστεύω ότι πρέπει να συζητήσουμε το εξή. Η Κομισιόν ε, δεν ε, το, Κοινοβούλιο δεν ε, πρέπει απλά να εγκρίνει κάποιες προτάσεις που έχουν γίνει στα κράτη-μέλη. Είμαστε εκλεγμένοι, συνομοθέτες και μας φαίνονται σαν να μην έχουμε καν εντολή. Έχουμε εντολή, μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι εάν ε, το υπαγορεύουν αυτό οι συνθήκες. μπορούμε να συζητάμε τα πράγματα εδώ στην ε, Επιτροπή μας, όπως άλλως θα κάνουμε σήμερα το απόγευμα αλλά έχω συχνά την ε, εντύπωση ότι ε, άλλοι μετακινούνται πολύ πιο δύσκολα από εμά. Επιτρέψτε μου να κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις ε, σχετικά με τα, με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και ο Λάμπερτ αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Όπως όλοι γνωρίζετε, Σημαντικά μέρη των ε, συμπερασμάτων αυτών αφορούν ε, την πολιτική συνοχής. Ελπίζω να μπορούμε να διαπραγματευτούμε εδώ, διότι φαντάζομαι το Συμβούλιο να λέει ότι μίλησαν τα αφεντικά, δεν έχουμε άλλη εντολή, δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Αλλά δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε συμβιβασμούς και ελπίζω να έχουμε και ουσιαστική υποστήριξη από την Κομισιόν. Και όσον αφορά αυτό που είπατε για ε, τους ε, προϋπολογισμούς ότι ε, αποτελεί απειλή το να για την περιφερειακή πολιτική το να κοιτάμε τα μεμονωμένα έτη μόνο. Από την άλλη όμως είναι απαραίτητο στις συζητήσεις να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό και για, να γίνει αυτό που μένει ακόμα δουλειά να γίνει. Για μένα δεν είναι πολύ σαφές εάν τα κράτη-μέλη γνωρίζουν ότι αν δεν φτάσουμε γρήγορα σε κοινό συμβιβασμό, τότε το Κοινοβούλιο ε, δεν έχει άλλη επιλογή από το να προχωρήσει σε πρώτη και δεύτερη ανάγνωση και έτσι ε, θα χάσουμε πολύ χρόνο. Δεν, δεν ξέρω αν τα κράτη-μέλη το γνωρίζουν αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω τους ε, συναδέλφους. Ε, ότι μπορεί στα κράτη-μέλη να πιστεύει ο κόσμος ότι κάποια στιγμή θα καταλήξουν σε κάποιο συμβιβασμό, ε, αλλά ε, δεν ισχύει αυτό. Πρέπει να γνωρίζουμε τι υπάρχει στη συνθήκη. Έχουμε συναπόφαση στην πολιτική συνοχή και γι' αυτό θα φροντίσουμε η διαδικασία της συναπόφασης πράγματι να είναι διαδικασία συναπόφασης και συνεργασίας. Θα χαρώ πολύ αν η Κομισιόν μας ε, στηρίξει στο θέμα αυτό και να κάνει θετικό lobbying, να το πούμε έτσι, στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ρωμόνα Μανέσκου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ. Δεν ε, θα κάνω εισαγωγικά σχόλια έτσι ώστε να αφήσω περισσότερο χρόνο στους συναδέλφους που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις και θα πράσω απευθείας στα ερωτήματα. Καταρχήν, πιστεύετε ότι ο προπολογισμό για την πολιτική συνοχή για την επόμενη περίοδο θα είναι αρκετός, ε, δηλαδή η πολιτική αυτή θα πετύχει τους στόχους που έχουμε θέσει στη Στρατηγική Ευρώπη 2020. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας να ξέρουμε πώς ε, θα καταναμηθεί αυτός ο προπολογισμός, πώς θα καταναμηθούν αυτά τα κονδύλια, έτσι όπως ε, ρώτησε ακριβώς ο κύριος ε, Φάνης Τελερόη. Δηλαδή θέλουμε να ξέρουμε ποια θα είναι τα νούμερα για κάθε πρόγραμμα, για κάθε κράτος. Όλα αυτά πρέπει να είναι σαφέστατα. Μια άλλη ερώτηση έχει να κάνει με το αποθεματικό επιδόσεων. Ποιο είναι, ποια είναι η δική σας άποψη και άποψη της Κομισιόν για το θέμα αυτό. Δηλαδή πώς θα καταναμηθεί το αποθεματικό αυτό. Αυτή είναι μία ακόμη πτυχή που θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη για μας να τη γνωρίζουμε στις διαπραγματεύσεις. Θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα πώς θα μοιάζει το μελλοντικό πρόγραμμα. Κατόπιν, σε σχέση με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα συμπεράσματα αναφέρουν ότι το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα συζητά κάθε δύο έτη την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής. Πώς ε, θεωρείτε εσείς ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο και πώς πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να οργανώσετε τη συζήτηση. Σκεφτήκατε να αντικατοπτριστεί αυτή η υποχρέωση σε ένα κανονισμό και τελευταία ερώτηση, επειδή ξεκινήσατε λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για τον Ισυντρία αναφερθήκατε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, ξέρουμε ότι έχει ληφθεί μια απόφαση στο Συμβούλιο ότι για δύο κράτη, για τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, η Κομισιόν ε, θα πρέπει να βρει πρακτικές λύσεις προκειμένου να μειώσει τον κίνδυνο των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση για την τρέχουσα περίοδο. Έχετε σκεφτεί ήδη κάποιες πιθανές λύσεις? Ξέρετε αν ε, θα μπορέσουν να βοηθήσουν ε, οι λύσεις αυτές στη Ρουμανία και στη Σλοβακία. ευχαριστώ. Ε, Εκεί που βρισκόμαστε τώρα για την έγκριση του Πολδίπ και λόγω της θέσης του Κοινοβουλίου Τη περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Καλό είναι που έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο. Ω προς το Ταμείο Συνοχής, η μεγαλύτερη απογοήτευσή μας, νομίζω ότι συμμερίζεται και η Κομισιόν, είναι ότι το μεγαλύτερο θύμα του Συμβουλίου είναι η πολιτική περιφερειακή συνεργασίας, η οποία περιορίζεται πια στο επίπεδο που είχε την προηγούμενη περίοδο. Ενώ εμείς και η Κομισιόν θέλαμε αύξηση. Ερωτώ λοιπόν, τι θα κάνουμε, τι θα κάνει η Κομισιόν για να μην θυσιαστεί αυτός ο στόχος. Δεύτερο θύμα είναι το πλαίσιο εκείνο των μεταβατικών περιφερειών που έχει και αυτό ροκανιστεί επειδή εμείς θελήσαμε λοιπόν να κρατηθούν δίκτυα, δίκτυα ασφαλείας για τις περιφέρειες που προέρχονται από το κοινό πλαίσιο τι θα μείνει από όλα αυτά για τις περιφέρειες μετάβασης λόγω των αυθαίρετων, μετά τις αυθαίρετες περικοπές. Απ' την άλλη, για τα διαδικαστικά τώρα, το Κοινοβούλιο τόνισε την αποφασιστικότητά του, δεν θα δεχτούμε τους αριθμούς που επέβαλε το Συμβούλιο και νομίζουμε ότι συμφωνούμε βασικά με την Κομισιόν, αλλά ότι σε αυτήν τη διαμάχη δεν νιώθουμε την Επιτροπή την Κομισιόν στο πλευρό μας. Πώς θα μπορούσε, τι θα μπορούσε να κάνει αύριο για να είναι λίγο πιο ενεργή ώστε να είναι αποδεκτό και από εμά το Πολδίπ. Για την Κούε Σαμαρτζή. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε που παρευρίσκεστε εδώ ενώπιόν μας και νομίζω ότι συνειδητοποιείται ότι η καλύτερη υποστήριξη της περιφερειακής πολιτικής ε, προέρχεται από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα από εδώ, από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δεν θα σας εκπλήξει το να σας πω ότι για μας ο κακός συμβιβασμός του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι απαράδεκτος. Πρόκειται για έναν απαράδεκτο συμβιβασμό, καθώς ε, στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισάγει τη λιτότητα που έχει δηλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο. Και με τον τρόπο αυτό δεν πρόκειται να ενισχύσουμε την πολιτική αλληλεγγύης που επιβάλλεται όλο ένα και περισσότερο για να βγούμε από την κρίση. Να σας πω ότι με εξέπληξαν τα συμπεράσματα ενός ερευνητικού κέντρου, αλλά τελικά έχουμε καταντήσει να διαβάζουμε τα συμπεράσματα ενός ερευνητικού κέντρου, γιατί δεν υπάρχουν πληροφορίες που να προέρχονται από την Κομισιόν, που να μας λένε ότι χώρες που θα χάσουν περισσότερο από την ισχύ του στο Συμβούλιο η Ελλάδα μείον 3%, η Ισπανία μείον 23% κτλ. Δηλαδή οι χώρες που ήδη πληρώνουν περισσότερο την κρίση και σε σχέση με όσο είπε ο Συνάδελφο Βανίστελ Ρόι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να τοποθετηθεί επ' αυτόν, αλλά δεν μπορεί να τοποθετηθεί παρά αν, ε, μόνο αν υπάρχει διαφάνεια. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώ είναι δυνατόν να γνωμοδοτήσουμε επί των αποφάσεων του Συμβουλίου, ενώ σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει παράσχει κανέναν υπολογισμό για την ένα κράτο και αναπεριφέρεια σύμφωνα με τους ε, κανόνες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και χωρίς αυτούς τους υπολογισμούς ε, πραγματικά μας είναι αδύνατο να αποφανθούμε. Σας ζητώ λοιπόν σήμερα να μας χορηγήσετε αυτές ε, τις πληροφορίες, αυτά τα αριθμητικά στοιχεία, τα πολύ συγκεκριμένα, το έκαναμε μια πρώτη φορά και το ξαναζητώ σήμερα. Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να πω. Βρισκόμαστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο, κατά κάποιο τρόπο χτίζουμε την ομολογία των ευρωπαϊκών θεσμών σε αυτό το νέο πλαίσιο διακυβέρνησης που προκύπτει από την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας και για πρώτη φορά θέτουμε σε εφαρμογή τη συναπόφαση. Και βλέπετε πόσες δυσκολίες ανακύπτουν στις διαπραγματεύσεις επίπεδο τριμερούς διαλόγου. Και έχουμε την εντύπωση πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επί σημείων που αφορούν την πολιτική συνοχή έχει ξεπεράσει τα δικαιώματά του και ότι στον τριμερή διάλογο κατά κάποιο τρόπο βρισκόμαστε πρώτοι τελεσμένων. Προσωπικά και νομίζω ότι θα πρέπει και νομικά να σταθούμε στο σημείο αυτό. Πιστεύω ότι κάποιοι κανόνες της συνθήκης έχουν παραβιαστεί. Και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει και αντικείμενο αντιδικίας. Ακούσαμε τι είπε και η Κωνστάς για το σημείο αυτό. Δεν είναι φυσιολογικό οι κανόνες της συναπόφασης να μην γίνονται απόλυτα σεβαστοί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να τηθεί πρωτοτελεσμένο, διαφορετικά οι τριμερείς διάλογοι δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαζίν και τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τον Επίτροπο να απαντήσει στους συντονιστές. Ειλικρινά Νομίζω ότι ο συνεχής τριμερής διάλογος ε, αποτελεί μια παιδαγωγική διαδικασία. Ε, να δείξει στο Συμβούλιο ότι το Κοινοβούλιο έχει ενισχυμένο ρόλο. Και μπορώ να συμφωνήσω με αυτά που είπε η Κωνσταντσα και άλλοι σχετικά με την επιτάχυνση. Συμβάλλουμε όπως μπορούμε, διότι και εμείς και εμάς μας ενδιαφέρει το θέμα και αυτό το έχω πει επανειλημμένα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να παραμείνει ως έχει η παρούσα αρχιτεκτονική ε, ακόμα και όταν μιλάμε για περικοπές και όταν φτάσουμε στο θέμα αν μπορούμε να ε, είμαστε ικανοποιημένοι με τις περικοπές. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι διότι ως Κομισιόν το 2011 υποβάλαμε πρόταση και η πρόταση αυτή ε, ήταν ήδη συμβιβασμός από την πλευρά μας. Και ε, βλέπαμε τι ήθελε το Κοινοβούλιο, βλέπαμε και τι έλεγαν ε, οι ε, καθαροί συνεισφορείς. Το Συμβούλιο έχει κινηθεί προς την κατεύθυνση των καθαρών συνεισφορέων, αλλά η Κομισιόν δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένη με κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα δούμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ο κύριος Αλφονσί αναφέρθηκε στην εδαφική συνεργασία. Παρακαλώ εδώ για τη συνεργασία σας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Να τονιστεί το θέμα αυτό, διότι σε σύγκριση με άλλα μέρη του προϋπολογισμού στην πολιτική συνοχής, δεν είναι σημαντικό όσον αφορά τα ποσά, αλλά είναι σημαντικό όσον αφορά το περιεχόμενο. Και με μια οικονομική αύξηση μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Όσον αφορά τις μεταβατικές περιφέρειες, και εδώ περιμέναμε περισσότερα, αλλά είναι σημαντικό το ότι υπάρχει η κατηγορία αυτή, είπαμε ότι ισχύουν αυτά για την παρούσα περίοδο, θα πρέπει να δούμε τι αποτελέσματα είχαμε, αλλά υπάρχουν οι μεταβατικές περιφέρειες και... και κατά την ε, κατανομή υπολογίζονται ανάμεσα στις περισσότερο ή λιγότερο μειονεκτικές περιοχές. θα πρέπει επίσης ε, να τονίσουμε ότι η ε, κατανομή γίνεται αναχώρα. Η πρόταση ήταν 5%, το Συμβούλιο λέει 7%. Το 2019 τα ποσά αυτά θα μοιραστούν εντός του κάθε κράτους μέλους ε, με βάση το αν τότε θα έχουν πετύχει τους στόχους τους ή όχι. Σε κάποιες περιπτώσεις θα έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, σε, κάποιους άλλους, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όχι. Το θέμα λοιπόν είναι αν θα έχουμε θετική ή αρνητική αντίδραση ε, ανάλογα με τα αποτελέσματα των ε, μεμονωμένων προγραμμάτων το 2019. Όσον αφορά την αντίδραση σε διάφορες ε, οικονομικές ε, εξελίξεις ή εξελίξεις ε, που έχουν να κάνουν με την απασχόληση, θα πρέπει να στηριχτούμε σε στοιχεία που έχουμε από την περιφερειακή πολιτική. Και στο προσεχές χρονικό διάστημα έχουμε τη ρήτρα αναθεώρησης για το 2016 με κάποιες τροποποιήσεις στον τομέα της ε, πολιτικής ε, συνοχής ε, που να ανέρχονται σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ζητάμε λοιπόν από το Κοινοβούλιο ρήτρα αναθεώρησης για το σύνολο του προϋπολογισμού. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται να διακυβεύσει την ασφάλεια προγραμματισμού, αλλά θα πρέπει να υπάρξει ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη οι, ε, εξελίξεις ε, μέχρι τότε. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλή η πρωτοβουλία αυτή. Επίσης, ε, όσον αφορά την υποχρέωση λογοδοσίας ε, κάθε δύο χρόνια στο Συμβούλιο, Πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο η πολιτική συνοχή να συζητιέται στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Ε, το πρότυπο που έχουμε ακολουθήσει εδώ, όπου ε, λίγο πολύ όλα τα κράτη-μέλη συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή. Ε, πιστεύουμε ότι είναι καλό και θα συνεχίσουμε να το έχουμε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, δηλαδή να συζητάμε τα θέματα αυτά. Κάτι τέτοιο δείχνει ότι τα καταφέρνουμε να θέσουμε τα θέματα σε επίπεδο Συμβουλίου προς συζήτηση. Ε, όσον αφορά το ερώτημα για συγκεκριμένα στοιχεία, υπάρχουν υπολογισμοί των κρατών μελών. Στις περισσότερες περιπτώσεις ε, δεν απέχουν πολλοί υπολογισμοί αυτοί από τους δικούς μας. Είμαι κάπως επιφυλακτικός ε, να αναφέρομαι σε νούμερα, διότι τα πράγματα ακόμα ρέουν. Θέλουμε να επικεντρωθούμε στην ουσία. Ε, να μπορέσουμε να εγκρίνουμε τους ε, σχετικούς κανονισμούς. Φοβάμαι ότι αν ε, ήδη σε τούτο το στάδιο επικεντρωθούμε υπερβολικά στα νούμερα, ουσιαστικά δεν θα προσέξουμε τα ουσιώδη. Αυτή τη στιγμή περνάμε ακόμα από μια διαδικασία ζήμωσης. Αλλά νομίζω ότι και σε οριζόντιο επίπεδο Ε, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν επιτρέπεται και δεν θέλω να προδικάσω. Ε, έλαβα το μήνυμα ότι Ε, όλοι οι συμμετέχοντες ε, στο τριμερή διάλογο θα πρέπει να μετακινηθούν. Αυτό ε, ισχύει και για την Κομισιόν, το κατάλαβα. Νομίζω όμως ότι ήδη έχουμε μετακινηθεί σε πολλά σημεία, αλλά όπως και για το Κοινοβούλιο υπάρχουν και για την Κομισιόν κάποιοι τομείς στους οποίους δεν μπορούμε να μετακινηθούμε καθόλου. Αν κατάλαβα σωστά, δεν απέχουν πολύ οι θέσεις μας. Μεταξύ τους έχουμε ήδη δεχθεί ε, ε, ε, Έχουμε συμφωνήσει σχετικά με την θεματική συγκέντρωση, όπου να μην έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων όμως τα θέματα, ε, να αφήσουμε στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες να καθορίσουν τις προτεραιότητες. Αυτό εννοούσα, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην επίτευξη των στόχων του 2020. και εξαρτάται από το είδος της περιφέρειας ε, ε, αν θα απελευθερωθεί το από 20 έως 50% του προϋπολογισμού για κάποια έργα. Υπάρχει λοιπόν θεματική συγκέντρωση ε, υπάρχει η ελευθερία για τη χρήση των υπόλοιπων ε, πόρων, ε, αλλά υπάρχει και ένα κατόφλι το οποίο προβλέπεται στο πλαίσιο του, της θεματικής συγκέντρωσης. Παρακαλώ λοιπόν να καθορίσουμε και αυτά τα στοιχεία και να μην αποδυναμώσουμε περισσότερο την πρόταση. Με τις τέσσερις κατηγορίες καλύπτουν με εντός του ERDF τα απαραίτητα. Και παρόλα αυτά ε, επιτρέπουμε και κάποιο περιθώριο για άλλα μέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Τώρα 14 άτομα έχουν ζητήσει το λόγο και έχουμε 45 λεπτά. Να δώσουμε ένα λεπτό στον Επίτροπο για να απαντήσει στον καθένα σημαίνει ότι χρειάζεται ένα τέταρτο περίπου. Έτσι λοιπόν, μισή ώρα έχετε για να μιλήσετε. Αν μακρηγορήσετε πάνω από δύο λεπτά, δεν θα είναι δυνατό οι τελευταίοι στον κατάλογο να παίρνουν το λόγο. Σας παρακαλώ, σεβαστείτε τα δύο λεπτά λοιπόν. Η πρώτη μιλήτρια, κυρία Κασιέσκα. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με όσα λέτε. Αυτή η συμφωνία μεταξύ αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων είναι κάτι σωστό και επίσης αν θέλουμε να εργαστούμε βάσει ετήσιων προϋπολογισμών αυτό θα ενείχε τεράστιους κινδύνους. Δεν θα μας επέτρεπε να υλοποιηθούν τα προγράμματα ούτε θα είχαμε ασφαλή σχεδιασμό ασφαλή προγραμματισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και έχει το δικαίωμα να θέσει επιφυλάξεις και επιχειρήματα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξή. Όταν βλέπουμε ποια είναι η δημοσιονομική κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη και όταν δούμε κυρίως τι συμβαίνει με τους καθαρούς συνεισφέροντες, ε, θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα να αυξηθεί ο προπολογισμό στα πλαίσια του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου, κυρίως σε ό,τι αφορά στην αγροτική πολιτική και την εταφική συνεργασία. Θα ήθελα να δράξω την ε, ευκαιρία σήμερα καθώς περιβρίσκεστε εδώ να σας ε, αναφέρω πόσο μεγάλες ανησυχίες υπάρχουν ε, στην περιοχή από όπου προέρχομαι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διακόψει την πρικοδότηση για αυτή την περιοχή, την ορεινή περιοχή της Πολωνίας, στην Νότια Πολωνία, σε σχέση με κάποιες ατασταλίες που δεν έχουν αποδεικτεί όμως κάτι τέτοιο έχει τεράστιες αρνητικές συνέπειες για όλη την περιφέρεια. Το δικό μας Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει καμία πληροφορία σε σχέση με το ποια πρικοδότηση τίθεται ε, σε κίνδυνο είναι δυνατόν να ανασταλεί. Μήπως η Κομισιόν θα ξεκινήσει μια νομική διαδικασία για να διαλύσει ε, αυτές ε, τις αμφιβολίες, γιατί πραγματικά είναι πολύ αρνητικέ οι συνέπειες. Επόμενος ομιλητής, ευχαριστώ πολύ. Θα παρακολουθώ το χρόνο. When we get the numbers. Θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν το εξή. Στις 7 Φεβρουαρίου συζητήθηκε το θέμα, τώρα είμαστε στο δεύτερο μισό του Μαρτίου. Εμείς κάναμε την πρόγνωσή μας, αλλά είναι ανεπίσημη και έτσι δεν μπορούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις των εκλογέων μας. Δεύτερον, τι θα κάνετε με τις ολονύχτιες παρουσίες στην Επιτροπή Περιφερειών ιδιαίτερα, όχι εδώ. Τα τελευταία δώρα που κάνατε εκεί 12,8 δισεκατομμύρια. Το έχετε αλλάξει αυτό καθόλου. Γιατί αυτά τα χρήματα παραμένουν στην προσθήκη δύο αλλά μήπως αλλάξετε την προσέγγισή σας για τις μεταβατικές περιφέρειες ή τελικά θα τα βγάλετε από εκεί. Και τρίτον, τι θα γίνουν τα λεφτά. Τον Ιανουάριο δεν πληρώθηκε τίποτα από το Ταμείο Συνοχής και το Περιφερειακό Ταμείο ή σχεδόν τίποτα. Ακόμα και για το Κοινωνικό Ταμείο τον Ιανουάριο δεν έγιναν πληρωμές. Σας κατευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επόμενος παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Επιτροπή, και εγώ λυπάμαι που έχουμε λιγότερα χρήματα για την περιφερειακή πολιτική και για τη γεωργία. Θα ήθελα να σας ζητήσω τη γνώμη σας επί της πρότασης της πολωνικής κυβέρνησης που θα ήθελε να μεταφέρει κονδύλια από την ε, πολιτική ανάπτυξη της υπαίθρου προς ε, άλλες πολιτικές, προς άλλα μέσα, γιατί αυτός ο προϋπολογισμός πραγματικά μειώθηκε κατά 25%. Έχουμε λιγότερα χρήματα τώρα στην πολιτική συνοχής. Δεύτερον, ε, για το έλλειμμα, δεν φοβάστε ότι αυτό το έλλειμμα θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο και στην πολιτική συνοχή, ε, γιατί δεν είναι δυνατόν να μειωθούν ε, οι δαπάνε στο πλαίσιο της γεωργίας. Πρόκειται για δαπάνε που δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Επομένως, αυτό θα επηρεάσει σίγουρα και την πολιτική συνοχή. Ε, μια ακόμη ερώτηση για τα 3,5 δισεκατομμύρια προοικοδότησης που αναστάλησαν για την Πολωνία και αυτό σχετίζεται με κάποιες υποτιθέμενες ε, ατασταλίες. Η πολωνική κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα μπλοκαριστούν αυτά τα χρήματα γρήγορα και έστειλε εξηγήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και τα χρήματα δεν έρχονται. Πότε θα απομπλοκάρει αυτά τα κονδύλια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει την πρόθεση να το κάνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπο, κύριε Σάλβες. Εγώ στο επίπεδο το υπεροπολογισμό των κονδυλίων που έχω εγκριθεί, θα ήθελα να πω ότι η Κομισιόν δεν αποτελείται από κάποιους ανθρώπους που τους αρέσουν οι περιπέτειες, όμως ε, το να έχει ζητήσει ένα διαφορετικό ποσό και να ε, ε, δέχεται τελικά 36 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα για τις πιστώσεις πληρωμών, όλα αυτά αμφισβητούν τα πάντα τα κονδύλια κονδύλια μειώθηκαν ε, σε πάνω από 23% σε ό,τι αφορά τους τομείς της ανταγωνιστικότητας. Επίσης και στο τομείς συνοχής ε, έχουμε εκεί μείωση 8,4%. Έτσι λοιπόν ένα από τα προβλήματα της σημερινής κρίσης είναι ότι έχουμε λιγότερα κονδύλια από ό,τι στο προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Όμως ε, δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για κονδύλια. Έχετε δίκιο όμως μας ανησυχεί και το εξή. Η τελευταία αξιολόγηση της Τροϊκά λέει ότι θα έχει η Πορτογαλία έλλειμμα 6,6%. και στη δική μου περιφέρεια το έλλειμμα είναι 0,4% μόνο και αυτό το υπολόγισε ε, και το χρέος 19%. Έτσι λοιπόν πώς θα εφαρμόσουμε την μακροαναλογία των διαφορετικών ταμείων και πώς θα αντιμετωπίσουν όλα αυτά οι πολίτες στη δική μου περιφέρεια όταν δεν φταίνε για το τι συμβαίνει σε επίπεδο χώρας και όταν αυτός ο κανόνας δεν είναι καθόλου διαρθρωμένος με το Σύμφωνο σταθερότητα και Ανάπτυξης που ποινικοποιεί τη χώρα και τη δική και μου περιφέρεια ε, έμεσα και όταν ε, δεν υπάρχει κανένας ε, κανόνας διάρθρωσης και εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει κάποιους κανόνες διάρθρωσης με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και να υπάρχουν αντικειμενικοί κανόνες εφαρμογής έτσι ώστε να μην ποινικοποιούνται οι πολίτες οι οποίοι ούτως ή άλλως έχουν μια διαφορετική συμπεριφορά. Uh, uh, Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Βόγκαν. Όπως και εσείς ε, και άλλοι συνάδελφοι στην αίθουσα, απογοητεύτηκα όταν η Συνοδός αποφάσισε μείωση των αριθμητικών στοιχείων για την πολιτική συνοχής και πρόσεξα όλα αυτά τα δωράκια που δόθηκαν, ένα δισεκατομμύριο εδώ, ένα δισεκατομμύριο εκεί και φτάσαμε τελικά στο ποσό των 13 δισεκατομμύριων ευρώ. Όμως ε, τα κράτη-μέλη θα προσπαθήσουν φυσικά να προστατεύσουν τις φτωχές περιοχές και ενα κρατη κράτο-μέλος που δεν προσπάθησε να το κάνει αυτό ήταν δυστυχώ το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί όταν ε, δείτε αυτό τον κατάλογο των δώρων ε, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν προστατεύει τις φτωχότερες περιφέρειες. Ξέρω ότι δεν έχουμε επίσημα στοιχεία ακόμη και άλλοι το σχολίασαν αλλά ξέρω ότι η κυβέρνησή μου έκανε την δίκη του και η Ουαλία θα έχει μείωση πάνω από 400 ε, εκατομμυρίων ευρώ και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έκανε το δικό της υπολογισμό και κατέληξε σε ένα παρόμοιο αριθμητικό στοιχείο. Η πρώτη ερώτηση είναι πώς ε, γίνεται η κατανομή στον Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ αυτών των διάφορων περιοχών και δεύτερον εσείς μπορείτε να το επηρεάσετε αυτό γιατί μου φαίνεται ότι είναι πραγματικά παράλογο οι πιο φτωχές περιοχές στο Ηνωμένο Βασιλείου να έχουν τόσο μεγάλες περικοπές στα διεθνωτικά ταμεία έτσι λοιπόν θα ήταν πολύ χρήσιμο να έχουμε τη δική σας επιρροή εδώ. Και δεύτερη ερώτηση ε, για τη δική μας επιρροή στους κανονισμούς που συζητάμε. Νομίζω θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και κάτι εμείς. Υπάρχει μία πρόταση τα κράτη-μέλη να μετεβάσουν όχι 2% αλλά 4% μεταξύ των περιφερειών και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βοηθήσει τη Σκοτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Εσείς τι πιστεύετε για κάτι τέτοιο, θα υποστηρίζετε ένα μεγαλύτερο ποσοστό που να μπορούσε να μεταφερθεί μεταξύ των περιφερειών. Ευχαριστώ. Ε, Άλλη μια ερώτηση, κυρία Ερικόνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχω τρεις ερωτήσεις να σας κάνω και σας ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Ελπίζω να μπορέσετε και να μου απαντήσετε. Μία ερώτηση έχει να κάνει με τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Η Κωνσταντς ρώτησε γιατί ανέκυψε εκ νέου αυτό το θέμα στον Συμβούλιο του Φεβρουαρίου. Και θα ήθελα να μου πείτε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και ποια είναι η θέση της Κομισιόν. Και αν ε, τελικά η μακροοικονομική αιρεσιμότητα, η πολλαπλή συμμόρφωση γίνει ε, αποδεκτή, πώς θα επηρεάσει την κατανομή των κονδυλίων. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με μια είδηση που εμφανίστηκε στον τύπο την περασμένη εβδομάδα και έχει να κάνει ότι υπάρχουν 50 δισεκατομμύρια από τα μία συνοχή ε, και διευθυντικά μία που δεν έχουν δαπανηθεί, ενώ ήδη... Ε, προσπαθούμε να θέσουμε σε εφαρμογή το σχέδιο δημιουργία της εργασία ε, και ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το τελευταίο ευρωμανόμετρο, αν η ανάπτυξή μα είναι 0,5%, μήπω η Κομισιόν ε, δεν θεωρεί ότι θα έπρεπε να τεθούν όλα αυτά σε εφαρμογή, ή υπάρχει άλλο τελικό προορισμό για αυτά τα κονδύλια και θέλουμε να περάσουμε ήδη στι περικοπέ για το επόμενο πολίτε δημοσιονομικό Και τρίτη ερώτηση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το 2012 διάφορα προγράμματα δεν ε, μπόρεσαν να καλυφθούν. Πώς η Κομισιόν ε, θα εγγυθεί ότι δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή το 2013 όλα τα προγράμματα τελικά να μπορέσουν να υλοποιηθούν όσα έχουν εγκριθεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μαρία. Επίτροπε έχετε ένα λεπτό ανά άτομο, τουλάχιστον 7 λεπτά δηλαδή. Ε, να ε, απαντήσω μαζί στην πρώτη και τελευταία ερώτηση. Από ότι κατάλαβα το θέμα αυτό είναι και μέρος των συζητήσεων για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να ε, αποφασίσουμε για έναν συμπληρωματικό προϋπολογισμό 12 δισεκατομμυρίων. την Άνοιξη προβλέψαμε 12 δισεκατομμύρια για ανοιχτές πληρωμές, να περάσουν δηλαδή στο παρόν έτος. Μιλάμε για μεταφορά από το 2011 στο 2012. Ε, έχει συσσωρευτεί λοιπόν εδώ πέρα ένας όγκος ε, πληρωμών που μεταβάζονται από το ένα έτος στο άλλο. Και έτσι φυσικά έχουμε πρόβλημα Ε, να κάνουμε κάποιες ε, πληρωμές. Αποτελεί λοιπόν ένα αίτημά μας για συμπληρωματικό προϋπολογισμό αυτό. διότι φυσικά μας ενδιαφέρει να υπάρχει ρευστότητα ε, εντός του κάθε έτους με βάση το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ήταν απαραίτητο να έρθουμε σε συμφωνία με ε, τα κράτη-μέλη ήδη κατά τις πρώτες ε, μειώσεις. Νομίζω ότι είχε ληφθεί υπόψη το θέμα αυτό. Όσον αφορά τις διάφορες ε, διακοπές, αυτό που είπα στον πολωνικό τύπο πριν κάποιες εβδομάδες. Τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε πάνω από 190 ε, διακοπές σε όλη την Ευρώπη. Νομίζω μόνο σε τέσσερις χώρες δεν το κάναμε αυτό. Από τις 190 αυτές διαδικασίες λοιπόν που επιτρέπεται να διαρκέσουν το πολύ ε, έξι μήνες, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ή τρεις αναστολές που είναι το επόμενο βήμα μέσα σε ένα εξάμεινο δηλαδή. Μπόρεσαν να λυθούν τα περισσότερα θέματα. Η Πολωνία έχει μερίδιο του προϋπολογισμού 20% ε, και έχει ε, μερίδιο στις ε, διακοπές αυτές 1 με 2%. Γενικά δηλαδή λειτουργούν καλά οι δομές της Πολωνίας. Αλλά βέβαια όταν υπάρχουν προβλήματα πρέπει να ενεργούμε εγκαίρως. Ε, δεν μπορώ να σας ε, δώσω πληροφορίες για τις ε, διάφορες επιμέρους υποθέσεις, αλλά οι συνεργάτες μου εργάζονται σκληρά με βάση τα έγγραφα που έχουν λάβει από τις διάφορες ε, κυβερνήσεις για να λύσουν τα θέματα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη ε, προϋποθετικότητα. Αυτό δεν επηρεάζει την κατανομή των πόρων, θεωρητικά μόνο, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις στο μέλλον. Κάτι τέτοιο δηλαδή θα μπορέσει να οδηγήσει σε διακοπή ή σε αναστολή των πληρωμών. Όσον αφορά τον συνάδελφο από την Ουαλία το εθνικό επίπεδο μπορεί να κάνει κατανομή των πόρων ε, ανάμεσα ε, σε ιδίου τύπου περιφέρειες, όχι όμως σε, διαφορετικές, ε, σε διαφορετικού τύπου περιφέρειες. Για παράδειγμα, στην έρευνα Μπορείτε όμως να είστε βέβαιος ότι κατά τις διαπραγματεύσεις θα εξετάσουμε την κατανομή εντός των κρατών μελών. Έχουμε το θέμα της Βρετανικής επιστροφής. Ε, το θέμα είναι πώς θα διασφαλιστεί αυτό να μεταβάσετε στις περιφέρειες. Υπάρχει λοιπόν ε, πάντα μια μεγάλη παρερμηνία. Δεν υπάρχει χρήμα που δεν απορροφάται. Υπάρχει το σύνολο των πόρων, το οποίο ήδη από την αρχή της περίοδου και σε ιδανική περίπτωση μάλιστα πράγματι στην αρχή της περίοδου. Μοιράζεται λοιπόν όχι μόνο μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, ε, αλλά και μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων. Και κατά τη διάρκεια των ετών Ε, παίρνουμε κάτι από αυτόν τον θεωρητικό λογαριασμό και το δίνουμε ε, σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ε, το επόμενο βήμα είναι όταν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αυτό και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες κοινοποιήσεις, τότε γίνονται οι πληρωμές. Τα 55 αυτά δις ήταν ένα ποσό που στο τέλος του 2011 δεν είχε μοιραστεί σε συγκεκριμένα, ε, ε, έργα, αλλά ε, είχε υπολογιστεί στον προϋπολογισμό των διαφόρων προγραμμάτων. Δεν είχε δηλαδή κατανεμηθεί στα επιμέρους έργα, αλλά όσον αφορά τα, τα προγράμματα είχε πράγματι μοιραστεί. Δεν υπάρχει χρήμα που δεν απορροφάται. Και θα ήθελα γι' αυτό να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι έχει καταρτιστεί προϋπολογισμός για τους πόρους και γι' αυτό μπορεί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και ανάλογα με τον κανόνα, νης είναι ένα, νης ε, ε, ε, ή δύο ή τρία χρόνια μετά το τέλος της αντίστοιχης περίοδου. Ε, δεν υπάρχει λοιπόν χρήμα που δεν να απορροφάτε του αντίον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πέντε ομιλητές έχουμε ακόμα. Παρακαλώ λοιπόν να σεβαστείτε τα δύο λεπτά. Ε, ο Πέτρο Λούχαν, ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ ιδιαίτερα ότι ο Επίτροπος ε, μιλάει ανοιχτά μαζί μας. Πρέπει να το εκτιμήσουμε αυτό. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μιλήσατε για τον κανόνα νη συν και είπατε ότι δεν θα συμβάλλει απαραίτητα σε μεγαλύτερη ε, δημοσιονομική αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, πολλές χώρες έχουν πρόβλημα όσον αφορά την απορρόφηση των πόρων. Δεν ε, είπατε όμως τι μπορείτε να βελτιώσετε ε, όσον αφορά το public acquisition μεγάλο ποσοστό των προβλημάτων οφείλεται ακριβώς σε αυτό το θέμα. Και δεν μας είπατε τι θα προτείνει η Κομισιόν και τι μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη ώστε να εφαρμόσουν ενιαία ομοιόμορφα μέτρα. Η δεύτερη ερώτηση ε, έχει να κάνει με, ε, την, ε, με, τον καλύτερο τρόπο δαπάνης των χρημάτων, το better spending. Έχετε κάνει συγκεκριμένη ανάλυση ανάλογα με το είδος των επενδύσεων. Δηλαδή, ποια χρήματα αποφέρουν την, αποδίδουν περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ερίκα Μάνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Θέλω να σας πω ότι έχω δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ γιατί υπερασπιστήκατε τον προπολογισμό για τις συνορικές περιοχές. Πιστεύω ότι εδώ ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης εμείς αγωνιστήκαμε έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη περιφερειακή συνεργασία και μάλιστα ζητήσαμε 7% του συνόλου του προπολογισμού. Όμως δυστυχώς το Συμβούλιο δεν είναι αρκετά πεπισμένο για τη σημασία αυτής της περιφερειακής συνεργασίας. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση και να επιμένουμε για αυτό το ζήτημα. Επίσης, σας υπενθυμίζω την ψηφοφορία της περασμένης εβδομάδας. Δυστυχώς δεν υπήρχαν αριθμητικά στοιχεία για αυτή την ε, συνεργασία, την περιφερειακή συνεργασία και λυπάμαι γι' αυτό. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να θίξω έχει να κάνει με τις ε, απομονωμένες περιοχές, ε, με χαμηλά ποσοστά πληθυσμού. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το τι κάνει το Συμβούλιο στο θέμα αυτό, γιατί αν υπάρχει μείωση των κονδυλίων θα υπάρχει πρόβλημα για αυτές τις περιοχές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα που είπαν ήδη άλλοι όπως τις δημόσιες προμήθειες. Αλλά να εκφράσω την ανησυχία μου για τις περικοπές στη γεωργία και στην πολιτική συνοχής. Επίσης ανησυχώ ιδιαίτερα για την διαμεθοριακή συνεργασία, γιατί και σε αυτήν θα γίνουν περικοπές. Καθώς και στην περιφερειακή συνεργασία. Δώσαμε ελπίδες στους εκλογείς μας και τώρα οι ελπίδες αυτές, οι προσδοκίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Είπατε ότι ίσως ο μόνος που υποστηρίζει τον κανόνα νη συν ο μόνος επίτροπος είστε εσείς. Μήπως θα μπορούσατε λοιπόν να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερο, είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα, είστε ο μόνος επίτροπος όντως. Επίσης είπατε ότι 45, 40% του νέου πολιτή θα χρησιμοποιηθούν για μετά το 2020. Αυτό αυτό με οθεί να σκεφτώ μήπως δεν χρειάζεται ήδη, μήπως ήδη από την αρχή δεν πάει για απόθεμα. Και γιατί να αρχίσει τόσο αργά το 20 μόνο και μετά. Εσείς ξέρετε καλύτερα τα πράγματα βέβαια ως προς τις εταιρικές συμφωνίες, την κατάσταση στα κράτη-μέλη κλπ. Αλλά είναι σαν να λέμε ότι όλα θα αρχίσουν με μεγάλη καθυστέρηση. Βάτσον. Ματσόνι, ματσόνι Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ε, ενδιαφέρουσα συζήτηση στην οποία συμμετέχουμε. Εσείς ε, εκφράσετε κάποιες ε, σκέψεις επί του προϋπολογισμού και μιλήσατε για αύξηση των πόρων, για την απασχόληση, την έρευνα και την ανάπτυξη και εκφράσατε τη θλίψη σας για την μείωση του προπολογισμού σε ό,τι αφορά τη γεωργία. Εγώ όμως θα να σας πω ότι πέρα από αυτό το αντιμενικό στοιχείο των πόρων για την πολιτική συνοχής, Υπάρχει μόνο ένα απόλυτο στοιχείο σε σχέση με τα κεφάλαια της καινοτομίας, της έρευνας και της απασχόλησης που επιβεβαιώνει αυτή την φωνή περί αύξηση Όμως στην πραγματικότητα η ανάλυση των δεδομένων μας οδηγεί στο να πούμε ότι όσα έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό δεν μας επιτρέπει να πετύχουμε τους στόχους ανάπτυξης και απασχόλησης που έχουν τεθεί από την ε, ίδια τη στρατηγική για το 2020 και αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό που δυστυχώς υποσκάπτει τις προπτικές ανάπτυξης. Ο κ. Κρέλ υπενθύμησε ότι εμεί ψηφίσαμε μια εντολή για την πολιτική συνοχή και εγώ θέλω να υπενθυμίσω ότι το Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα υιοθέτησε και ένα ψήφισμα σε σχέση με την απόφαση του Συμβουλίου για τον προπολογισμό. Εγώ πιστεύω ότι η θέση που εκφράζεται στα έγγραφα αυτά πρέπει να τις υπερασπιστούμε, τις θέσεις αυτές, όχι μόνο ε, επειδή υπάρχει λόγος ολοζωντής, αλλά επειδή είμαστε πεπισμένοι για το αποτέλεσμα που πετύχαμε, γιατί αποτελεί το αποτέλεσμα ε, μιας ε, εις βάθος δουλειάς. Και αν με επιτρέπετε θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Εσείς μιλήσατε ότι δεν ε, υπάρχει συνέχιση από τη μία στρατηγική στην άλλη και αυτό το πέρασμα χωρίς συνέχεια ε, θεωρείται ότι έχει να κάνει και με τη διάθεση των πόρων μεταξύ ε, των πόρων που έχουν δεσμευθεί και των πόρων ε, που έχουν δαπανηθεί για να καταλήξουμε σε μια δυνατότητα απεμπλοκής όταν ε, μιλάμε για ένα κράτος που δεν έχει κατορθώσει να δαπανίσει Δηλαδή, να αναφερθώ στην Ιταλία, δεν έχει κατορθώσει να δαπανίσει παραδείγματο χάρη του ε, πόρου για την επόμενη στρατηγική. Θα πρέπει να ποινικοποιηθεί η Ιταλία. Είναι ανοιχτή αυτή η συζήτηση. Σε ό,τι αφορά τη θεματική συγκέντρωση, συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Πολύ σωστά να διατηρήσουμε την οργάνωση για να υλοποιηθούν ε, οι δαπάνες όμως πιστεύω ότι είναι σημαντικό να σκεφτούμε και επί της ευελιξίας στο, στο πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι. Γιατί αυτή η έλλειψη ευελιξίας μας οδήγησε στον αποτύχει η Λισαβόνα του 2010, η στόχη της Λισαβόνας 2010 που είχε, οργανωθεί, που είχε οργανωθεί βάση της αρχής της συγκέντρωσης και μακροοικονομική ρεσιμότητα. Ο κύριος Ρέ μιλά για αναθεώρηση των κριτηρίων ε, που εμπνέουν το Σύμφωνο Σταθερότητας ε, και συγκεκριμένα σε σχέση με τις επενδύσεις. Εμείς σήμερα, ενώ η Κομισιόν κάνει αυτό το σημαντικό βήμα προς τα μπρος σε σχέση με την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας, επιδεινώνουμε ε, τη θέση μας σε σχέση με τις επενδύσεις που στηρίζουν την πολιτική συνοχή. Σε ποια είναι η δέσμευση της Κομισιόν σε σχέση με όλα αυτά? Ο κύριος Ουντιάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τη διαθεσιμότητά σας. Ε, μια ερώτηση εγώ θέλω να κάνω, όχι παρέμβαση, για να αφήσω και χρόνο να απαντήσετε. Η ερώτηση μου δεν αφορά τα αριθμητικά στοιχεία, αλλά τη διαδικασία. Και συγκεκριμένα το γενικό κανονισμό που εγκρίναμε και που ε, εντοπίζει την διαδρομή ε, ως μια ενάρετη διαδρομή για να έχουμε αποτελεσματικές ε, δαπάνες των κονδυλίων για να ξοδέψουμε πολιτισματικά το κονδύλιο. Πώς ξέρουμε ότι δεν θα υπάρχει εμπλοκή σε αυτό το θέμα στον τριμερή διάλογο και πώς ε, ξέρουμε ότι πολλές περιοχές ε, θα μπορέσουν ε, να συμμετέχουν σε αυτή τη σύμπραξη. Και θέλω να ρωτήσω, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση των άτυπων διαπραγματεύσεων με τα κράτη-μέλη Βλέπω ότι γνέφεται. Περιμένω την απάντηση, λοιπόν, δεν συνεχίζω. Ευχαριστώ. Ernst. Nee, das ist nicht. Doch, es ist es. Okay, Entschuldigung. Ja. Nein, Sie genommen. Kiri, Petrope. βρίσκω ότι ως Κομισιόν ε, κρατάτε αμυντική θέση και ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, στην Αυστρία θα συμφωνούσατε με προϋπολογισμό όπου ξεκινάτε ήδη με κάποιο ε, έλλειμμα το οποίο δεν καλύπτεται ούτε από ε, φορολογικά έσοδα, ούτε από κρατικά έσοδα, ούτε από ε, κάποιο δάνειο. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα κενό το οποίο δεν καλύπτεται. Και ε, απ' την άλλη ε, έχουμε ε, το δημοσιονομικό κανονισμό, ο οποίος μιλάει για μείωση των... Μιλάει για περικοπές. Η κατάσταση λοιπόν που αντιμετωπίζουμε τώρα, η κατάσταση αυτή απαιτεί από την Κομισιόν να πει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Αυτό θα ήθελα να δω από την Κομισιόν. επόμενη παρατήρηση. Έχετε κάποιον Ε, έχετε κάνει κάποιον ε, ε, υπολογισμό σχετικά με το τι θα σημάνουν αυτά τα 960 δισεκατομμύρια για την συνοχή ή στη χειρότερη περίπτωση 908 δισεκατομμύρια. όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στην συνοχή, στο σύνολό της. θα πρέπει να υπολογίσουμε τι θα γίνει και στην χειρότερη περίπτωση. και εγώ προέρχομαι από μεταβατική, περίοδο, μεταβατική περιφέρεια. και έχουμε σοβαρά προβλήματα. Τι θα πούμε στον κόσμο σχετικά με την όλη κατάσταση. Επίσης, ε, η εντολή του Συμβουλίου ε, ξεπεράστηκε διότι ζητήθηκαν περισσότερα. για τον προϋπολογισμό. Το Συμβούλιο έκανε πολύ περισσότερα από ό,τι του επιτρέπεται. Ε, ε, πρόκειται για παραβίαση της συνθήκης. Ε, τι θα κάνετε με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, Καρή Μαντέλη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, όπως ε, είπαν και οι συνάδελφοι, στην Ευρώπη αξίζει κάτι περισσότερο από έναν τέτοιο προϋπολογισμό να σας πω πόσο απογοητευμένοι είμαστε. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα μυρολατρείας κύριε Επίτροπε, καιρός είναι συλλογικά να οικοδομήσουμε το μέλλον όπως είπατε και εσείς και ιδιαίτερα για τους νέους. Πάρτε λοιπόν ένα κλειδί, η ενεργειακή μετάβαση. Είναι η μεγαλύτερη πρόοδος που μπορεί να γίνει σε αυτόν τον αιώνα και θα σηματοδοτήσει την αλλαγή. Μιλήσατε για την ανεργία. Όταν δούμε τι μπορεί να γίνει και ως προς αυτό για τις ανανεώσιμες πηγές, για την εξοικονόμηση, αποδοτικότητα της ενέργειας με τη γεωθερμία κτλ. Να, κοινωνικές, κοινωνικώς αποδεκτές λύσεις. Λοιπόν, για την ενεργειακή μετάβαση κύριε Επιτροπέ μου, πρέπει να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε σε μια φάση όπου αρχίζουν να σπανίζουν οι πρώτες ύλες, οι πόροι, οι ενεργειακοί πόροι, οι γνωστοί. Και άρα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πετύχουμε την μετάβαση από μία, σε μία ενέργεια χωρίς διοξίδιο. Εγώ φοβάμαι πολύ ότι το Συμβούλιο θα αποδυναμώσει στη θεματική συγκέντρωση αυτά τα θέματα. Και βλέπουμε ήδη ότι το Συμβούλιο θέλει να επιβάλλει τα δικά του θέματα με εκβιασμό, ιδιαίτερα μέσω του λεγόμενου μηχανισμού διασύνδεσης. Για να καταλήξουμε λοιπόν κύριε Επίτροπέ μου στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των δυνατοτήτων μας πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τα εργαλεία ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Ελπίζω να πείσετε και τα κράτη-μέλη, να εξηγήσετε δηλαδή πόσο καλά είναι τα IT. Ε Έχετε μπροστά σας πεδίο δόξης. Τώρα πρέπει να γίνει αλλαγή, όχι σε δύο χρόνια ούτε σε τρία. Τώρα, τώρα παίζεται το πράγμα. Σε εσά υπολογίζω λοιπόν για να εκμεταλλευτείτε αυτή τη νέα δυναμική. Κυρία Φεραγκούτ, ε, κοιτάξτε, εγώ προέρχομαι τις Βαλεαρίδες και ιστορικά όλα τα νησιά το έχουν ζητήσει. Εμείς ε, δεν συμφωνούμε με το όριο του 150 χιλιόμετρων για τη διασυνορική συνεργασία δεν κατανοώ γιατί το όριο αυτό, δεν καταλαβαίνω γιατί οι Βελαιορίδες δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το ταμείο, που θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και έχει υποστηρίξει πολύ καλά project ε, και επίσης ε, οι συνθήκες λέ, μιλάνε για οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Ε, η συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρεται στο θέμα αυτό, παρόλα αυτά δυστυχώς συνεχίζουμε να υφιστάμεθα διάκριση και η έκθεση του Κοινοβουλίου έλεγε ότι θα έπρεπε να μην ισχύει αυτό το όριο απόστασης ε, για τα νησιά. Δεν καταλαβαίνω γιατί το Συμβούλιο συνεχίζει να διατηρεί το όριο αυτό. Η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία έχουν ζητήσει την εξάλληψη αυτού του όριου για τα νησιά. Η Φιλανδία πιστεύετε ότι θα κάνει, μάλλον Έχετε σκοπό να κάνετε κάτι για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, Κάτριν Μπέρντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί δεν έχουμε χρόνο. Οπότε καταλάβει η Κομισιόν έχει μια μυθοδολογία να διασφαλίσει ότι τα κρατη δεν έχουν τη μόνη ευθύνη για την κατανομή των πόρων στις περιφέρειες. Και αναρωτιέμαι αν η Κομισιόν μπορεί να διασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη έχουν την ευελιξία να κατανείμουν τα κονδύλια σύμφωνα με τις δικές σας προτεραιότητες. Ακούσαμε αριθμητικά στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυκλοφορούν πάρα πολλά νούμερα στον τύπο. Η αυξανόμενη χρηματοδότηση των περιφερειών ανάλογα με τον πληθυσμό και ε, κάποιες περιοχές με πολύ πληθυσμό βρίσκονται εκτός. Έτσι σκοπεύετε να εξοδεύσετε τα χρήματα και αν όχι, πώς θα ελέγξετε Δηλαδή, πώς θα προσδώσετε ευελιξία μεν και πώς θα διατηρήσετε και τον έλεγχο σε σχέση με τη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ, κύριο Επίτροπο τώρα και τις τελικές παρατηρήσεις. Να μας πείσετε, τελευταία σα ευκαιρία. Ίσως να ξανακάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τις πληρωμές. που υπάρχει στην ε, απόφαση ε, των ε, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Στο διάστημα 2007 έως 2020 προβλέπονται πληρωμές 908 δισεκατομμύριων. Αλλά συνολικά στα 7 χρόνια μπορούμε να διαθέσουμε κάτι λιγότερο από 960 δισεκατομμύρια το ποσό που ξεπερνά τα 908 μπορεί να πληρωθεί τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι η σχέση ανάμεσα σε αυτά τα ποσά. Πριν λοιπόν που μίλησα για το 40% ουσιαστικά Όσον αφορά τα ποσά, έχουμε de facto ε, ένα διάστημα 10 ετών. Και θα πρέπει να έχουμε κατά νου πώς εφαρμόζονται τα προγράμματα και προς το τέλος προς το τέλος της περίοδου αυτής ε, αυξάνεται η ολοκλήρωση των, ε, των ε, έργων, οπότε θα πρέπει να πληρωθούν περισσότερα ποσά. Στο τέλος δηλαδή της περίοδου αυτής γίνονται περισσότερο πληρωμές από ό,τι στην αρχή και γι' αυτό μιλώ για δεκαετία. Είναι συντηρητικός ο υπολογισμός μας που λέει ότι το 40% του προπολογισμού μας, ε, ε, του προϋπολογισμού μας εκείνο το χρονικό διάστημα θα πρέπει να πληρωθεί. Αλλά μπορούν τα κράτη-μέλη να συντομεύσουν την ε, διαδικασία, είναι προς συμφέρον τους. Με τον κανόνα νη συν το ότι η πίεση να ολοκληρωθούν τα προγράμματα μειώνεται. θα ήταν σαν να υποθέτουμε ότι μετά το 2020 θα υπάρχουν νέα προγράμματα. Ε, το αντίθετο συμβαίνει. Ε, όταν ολοκληρώνονται προγράμματα μπορούν να ε, ε, ξεκινήσουν καινούρια. Όταν λοιπόν έχουμε διάστημα επικάλυψης τρία χρόνια υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι και Γι' αυτό δεν είμαστε ενθουσιασμένοι με το θέμα αυτό. Η κυρία Μανέσκου ήδη έφυγε. Ε, αλλά για τη Ρουμανία, τη Σλοβακία κλπ. θα πρέπει να βρούμε μια δυνατότητα. Εξετάζουμε τι μπορεί να γίνει ώστε να ανταποκριθούμε στις επιθυμίες που έχουν εκφραστεί. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας δώσω κάποιο αποτέλεσμα, διότι εξετάζουμε ακόμα την κατάσταση. Θέλουμε να αποφύγουμε τροποποίηση των κανονισμών, ώστε να μπορούμε να περάσουμε στην εφαρμογή. Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, αυτό είναι τρέχον θέμα. Έχουμε κάποια μέτρα απλοποίησης, αλλά είναι σημαντικό και νομίζω ότι σημαίνει αυτό στη Ρουμανία, αλλά δεν είμαι απόλυτα ενημερωμένο. Να ε, χρησιμοποιούνται ενιαία διεθνή έντυπα για τους δημόσιους διαγωνισμούς ε, και όσον αφορά την ε, ποιότητα των επενδύσεων, την καλύτερη απόδοση των χρημάτων. Δεν μπορώ να σας δώσω εδώ μία σύντομη απάντηση. Μπορώ να σας πω μόνο ότι μας ενδιαφέρει το ποσοστό των ε, χρηματοπιστωτικών μέσων να αυξηθεί σημαντικά στο επόμενο χρονικό διάστημα, ε, στο, μάλλον θα ανέρχεται το ποσό στα 10 δισεκατομμύρια. Αλλά βέβαια όλα εξαρτώνται από τις δυνατότητες που υπάρχουν, ε, από τις συνθήκες που θα επικρατούν στο προσεχές χρονικό διάστημα. διότι ε, έτσι έχουμε τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα μόχλευσης. Υπάρχουν ε, όμως ε, συνθήκες που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν διαφορετικά benchmarks, διαφορετικά σημεία αναφοράς τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, τα οποία είναι διαφορετικά για κάθε χώρα. Αλλά θέλουμε να αυξήσουμε την ποιότητα της πολιτικής. Ευχαριστώ όσους αναφέρθηκαν στην εδαφική συνεργασία. Σημειώνω ότι το Κοινοβούλιο ε, πολύ σοφά δεν έχει προτείνει συγκεκριμένα νούμερα. Κατάρτιση του προϋπολογισμού και ταμεία. Αν η στρατηγική της ε, Λισαβόνας ε, δεν ε, πέτυχε, τουλάχιστον μάθαμε διάφορα πράγματα από αυτό. Δεν μπορούμε ταυτόχρονα να διασπάσουμε τους στόχους για τα διάφορα κράτη κατευθείαν σε στόχους για τις περιφέρειες και σε τοπικό επίπεδο. Προφανώς για πολλές χώρες και περιφέρειες δεν ήταν αρκετά φιλόδοξη η στρατηγική. Ε, όπως ε, είπα, η επελιξία δεν επιτρέπεται να παρερμηνευτεί. στο πλαίσιο των ε, συνθήκων που δεσπόζουν επιτόπου θα πρέπει να βρεθεί μία λύση στα μέτρα της κάθε περιφέρειας. Και όταν μιλάμε για το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και την σχέση μεταξύ τους, ξέρουμε ότι έχουμε το Κοινοβούλιο στο πλευρό μας ε, όπως έχουμε πει η κατάσταση που επικρατεί στο κάθε κράτο μέλος είναι διαφορετική αλλά μπορεί το Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με το θέμα αυτό ώστε στις ε, διάφορες χώρες ε, να έχουμε διαφορετικές διαδικασίες σε πολλές χώρες, σε τοπικό επίπεδο. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου δεξιότητες και ακριβώς για αυτό το λόγο δεν έχουν το απαραίτητο διοικητικό δυναμικό ώστε να εφαρμόσουν τέτοια προγράμματα. Υπάρχουν ε, διάφορες προϋποθέσεις ε, και ως ε, περιφερειακός πολιτικός, κάποιος που προέρχεται από το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, θέλω μια λογική ανάπτυξη δεξιοτήτων, ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο, εκεί όπου έχει νόημα κάτι τέτοιο. Θέλουμε φυσικά και καλύτερη χρήση των ε, πόρων σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχουν ε, καταρχήν κανόνες για κάτι τέτοιο, τους οποίους ε, δεν μπορούν να παρακάμψουν τα κράτη-μέλη εφόσον έχουν συμφωνηθεί. Και σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς θα δαπανηθούν οι πόροι. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών βρίσκονται σε καλό δρόμο και στις ε, χώρες όπως η Ιταλία, όπου σε πολιτικό επίπεδο είχαμε διάφορα, ε, διάφορες διακοπές. Σε διοικητικό επίπεδο τα πράγματα προχωράνε καλά. Η... Ωστόσο, ε, οι ανισότητες ανάμεσα στις περιφέρειες δεν βοηθάνε τις διαπραγματεύσεις, αλλά αυτή τη στιγμή πάνε καλά τα πράγματα. Και δεν νομίζω ότι έχω κρύψει τις θέσεις μου. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι ε, δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε χρέη ε, και το 40% του προϋπολογισμού ε, ε, επανέρχεται στα κράτη-μέλη για διάφορες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες. Εάν λοιπόν μειωθεί ο προϋπολογισμός θα είναι λιγότερα και τα χρήματα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τα 150 χιλιόμετρα. Υπάρχουν συζητήσεις. Η Κομισιόν θα επιδείξει ευελιξία, αλλά θα πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στην ε, άμεση συνεργασία ε, και το να συμμετέχει κανείς σε ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα. Οι βαλερίδες ε, μπορεί να έχουν εδώ πέρα διάφορες δυνατότητες, αλλά θα πρέπει να υποβληθούν σχετικές προτάσεις και να αναλυθούν οι απαραίτητες ευθύνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. φαντάζομαι ότι θα έχουμε και στο μέλλον συναντήσεις. Ε, οι επόμενοι μήνες ε, θα είναι αποφασιστική σημασίας. Και στα περισσότερα θέματα νομίζω ότι η Κομισιόν ε, συμφωνεί με το Κοινοβούλιο και οι δύο ενδιαφερόμαστε να βρούμε λύσεις. Και άλλωστε έχουμε και κοινό συμφέρον να έχουμε καλό προϋπολογισμό σχετικά γρήγορα και σύντομα να μπορέσουμε να, να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία προς συμφέρον των πολιτών μας. ευχαριστώ πολύ. Thank you, Don't forget that you are... Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Όποτε θέλετε να μας μιλήσετε, μην ξεχνάτε ότι είστε πρόσδεκτος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ετοιμότητά σας και την ε, πρόθεσή σας να απαντήσετε όλες αυτές τις ερωτήσεις ε, και φυσικά βασιζόμαστε στην υποστήριξή σας για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Στις 3.30 θα ξανασυναντηθούμε για να συζητήσουμε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης της Ρουμανίας και τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ρουμανίας για να συζητήσουμε το μέλλον της πολιτικής στη Ρουμανία.